Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Platz zu nehmen. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ. Έχουμε κάποια σχετική πίεση χρόνου. Νομίζω ότι έχετε εγκρίνει τη μέση διάταξη. Αν έχετε κάποια αντίρρηση, πέστε μου τώρα. Να σας κοινοποιήσω το γεγονός ότι η Υπηρεσία Εξωτερικών, Εξωτερικής Δράσης θέλει να λάβει το λόγο στην ε, περίπτωση της Σερβίας λόγω της, ε, λόγω της ε, σύλληψης τους, εντάλματος κατά του Ραμού Σαλντίνα, του πρώην πρόεδρου του Κοσφοπεδίου. Και θέλω εδώ να εκφράσω την, επίσης τη λύπη μου, την θλίψη μου για την θανάτωση, για, τον, για τη δολοφονία μάλλον Ισραηλινών στρατιωτών στην Ιερουσαλήμ από μια τρομοκρατική ενέργεια. Εμείς θα πάμε στην Ιερουσαλήμ με μια αντιπροσωπεία μάλλον είχαμε πάει με μια αντιπροσωπεία της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων κοντά στην Κνεσέτ και ήμασταν πολύ κοντά στο σημείο που μετά από μερικές μέρες έγινε αυτή η τρομερή τρομοκρατική ενέργεια. Πιστεύω λοιπόν ότι και εσείς θα συμφωνήσετε να εκφράσω προς τους συναδέλφους μας στην Κνεσέτ την ε, συμπαράστασή μας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. τα πρακτικά θα ακολουθήσουμε και εκεί την ε, πάγια διαδικασία. Θα εγκριθούν εάν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση και έρχομαι τώρα στο θέμα της Δυτικής Σαχάρας. Ο κύριος Νίκολας Βέσκο, Βέσκο ο οποίος είναι ο διευθύνων για την ε, Μέση Ανατολή και την Νότια Αφρική, θα μας ε, δώσει την άποψη της ε, Ευρωπαϊκής ε, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης μετά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την προσφυγή του μετόπου Πολυσάριου. Έχετε το λόγο κύριε Westcott. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά είμαι και πάλι μαζί σας με την Επιτροπή ΑΦΕΤ. Καλή χρονιά για αυτούς που δεν έχω δει ακόμα. Στις 20 Δεκεμβρίου, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε ένα συμπέρασμα για την περίπτωση για την ε, προσφυγή του, Συμβουλίου... Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εναντίον της ε, απόφασης που είχε κάνει το πρωτοδικείο σε σχέση με την απόφαση του Συμβουλίου για τις αγροτικές επιδοτήσει στην περίπτωση της Δυτικής Σαχάρας. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η διαδικασία αυτή με το να εγκρίνει την απόφαση του, την προσφυγή του Συμβουλίου και να ακυρώσει την απόφαση του Πρωτοδικίου στις 15 Δεκεμβρίου επικυρώνεται. Το αποτέλεσμα είναι ότι η απόφαση του Συμβουλίου που οδηγεί στη σύναψη της αγροτικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκο παραμένει ισχύ και δεν έχει ακυρωθεί ούτε καν εν μέρη όπως είχε αποφασιστεί καταρχήν από το πρώτο δικαστικό επίπεδο. Πρέπει όμως να υπογραμμίσω ότι όταν έγινε αυτή η προσφυγή από την πλευρά του Συμβουλίου και αυτό έγινε με ομόφωνη θέση του Συμβουλίου με την υποστήριξη των κρατών μελών κάποια από τα κρατημέλη παρενέβησαν ω ε, διάδικοι και στη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου, υποστηριζοντας τα επιχειρήματα που παρουσίασε η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου. Αμέσως μετά την ε, απόφαση του Συμβουλίου, την ίδια μέρα, 21 Δεκεμβρίου, εξεδόθη μια κοινή δήλωση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Μαρόκου και από την ε, ύπατη εκπρόσωπο, κύριε Μογκερίν, όπου και οι δύο πλευρές καταγράφουν και λαμβάνουν γνώση της απόφασης του δικαστηρίου ε, έχουν λαμβάνουν γνώση του γεγονότος ότι θεωρήθηκε μη παραδεκτή η προσφυγή η περίπτωση αυτή και είναι έτοιμοι να συνεργαστούν για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή αυτής της απόφασης στο πλαίσιο της ε, προνομιακής εταιρικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκο. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει και την στρατηγική φύση της σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μαρόκο που παραμένει πάρα πολύ σημαντική και για τι δύο πλευρέ. Το Μάροκο εξακολουθεί να είναι ένα κέριο εταίρο στη νότια μα γειτονία, με τον οποίο έχουμε δημιουργήσει μια πάρα πολύ σημαντική και πολύτιμη εταιρική σχέση τα τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προσιλωμένη στην ενίσχυση αυτής της σχέση Θα εξετάσουμε τη δυνατότητα ε, επισκέψεων σε υψηλό επίπεδο και από τις δύο πλευρές για να επαναληφθούν οι σχέσεις συνεργασίας στους τομείς όπου είχε ανασταλεί αυτή η συνεργασία. Για την ίδια την απόφαση, η οποία φυσικά είναι δεσμευτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της, βρισκόμαστε στη διαδικασία του να εξετάσουμε τις πλήρεις συνέπειες αυτής της, ε, συμφωνία, της απόφασης, τις νομικές συνέπειες. Αυτή η ανάλυση θα απαιτήσει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των νομικών υπηρεσιών της Κομισιόν του Συμβουλίου της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Αυτή η διαδικασία είναι εν εξέλιξη. Αλλά παραμένουμε και σε στενή επαφή με τις αρχές του Μαρόκου, οι οποίες ε, φυσικά και αυτές ενδιαφέρονται για αυτή την απόφαση και που είναι οι προνομιακοί μας συνομιλητές για το θέμα αυτό. Έχουν λάβει χώρα επαφές σε υψηλό επίπεδο καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης της προσφυγής και 21 Δεκεμβρίου, ο κύριος Μπελιάρ, ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν εκεί για να υποβεί τη σημασία που έχει εκεί για το Μαρόκο και για τα κράτη-μέλη αυτή η υπόθεση. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν. Η απόφαση λοιπόν για τη συνεργασία παραμένει. Δεν έχει γίνει δεχτή η προσφυγή του Πολυσάριου και αυτή είναι η κατάσταση. Θέλει κάποιος να λάβει το λόγο. Штетина. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμε κύριε Διευθυντά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το Μαρόκο αποτελεί σημαντικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τους τελευταίους μήνες ε, το είδαμε αυτό επανειλημμένα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και θέματα των προσφύγων, το ρόλο που έπαιξε το Μαρόκο σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες. Και να σας υπενθυμίσω και το εξή, Ο Μοχάμετ, ο 16 ο βασιλιάς του Μαρόκο, ήδη πέρσι δήλωσε ότι το Μαρόκο είναι μία από τις πρώτες χώρες ε, του Νότου που ακολουθούν μια αυθεντική αλληλέγγυα πολιτική για τους πρόσφυγες της υποσαχαρής Αφρικής και να σας πω ότι από την πολιτική μου εμπειρία γνωρίζω ότι η δεύτερη φάση ενσωμάτωσης των μεταναστών επίσης είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει και θα πρέπει να ακολουθήσει την πρώτη φάση, η οποία ξεκίνησε το 2014. Και οι δύο οι φάσεις αυτές ε, περιλαμβάνουν ε, την κάλυψη 25.000 25.000 μεταναστών προσφύγων από την ε, υποσαχάρια περιοχή. Δεν μπορώ παρά να επενέσω λοιπόν τις προσπάθειες αυτές του Μαρόκο. Αλλά το θέμα είναι τι θα γίνει και για την ενσωμάτωση των ανθρώπων αυτών. Πώς θα ενσωματωθούν στην ε, κοινωνία του Μαρόκο. Η ενσωμάτωση, ξέρετε, 50.000 ε, ατόμων δεν είναι μικρό πράγμα. Μικρό πράγματα. Ε, ξέρετε. Ότι το Μαρόκο λοιπόν θέλει να ενσωματώσει 50.000 άτομα. Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί και πώς θα το πετύχει το Μαρόκο αυτό. Συνάδελφε, λέει ο Πρόεδρος. Θα γίνουν αντιπαθή και πάλι και τελειώνει η θητεία μου, αλλά δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Έχουμε ακόμα δέκα άτομα που ζητούν το λόγο και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει όλοι να περιοριστείτε στο ένα λεπτό. Συμφωνείτε? Συμφωνείτε. Ο κ. Πανιού. Κύριε Πρόεδρε, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θέτει τέλος ε, ε, στις απαιτήσει και των φίλων ε, Μαροκινών και πιστεύω ότι η ανάκτηση μιας υγιούς σχέσης με το Μαρόκο θα πρέπει να γίνει, γίνονται διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή επιτάπητος με τον ΟΗΕ. Ο κύριος Westcott το ανέφερε, το θέμα είναι πώς προβλέπει να βοηθήσει ή να συνοδεύσει το νέο Γενικό Γραμματέα Γκουτιέρες σε αυτό το έργο. Δεύτερον, θα πρέπει να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε ώστε να ε, δούμε ακριβώς ε, και να αντιμετωπίσουμε τις βασικές προκλήσεις με το Μαρόκο, που είναι ο βασικός μας εταίρος σε θέματα μετανάστευσης, αλλά επίσης την ε, περιφερειακή σταθερότητα και την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών αλλαγών. Ποια μέτρα λαμβάνετε για να ενισχύσετε αυτή την εταιρική σχέση τώρα που έχει περάσει αυτό το, η περίοδος παγώματος αυτού του ε, νομικού επεισοδίου. Spoštovani, imamo Evropskega Έχουμε μια απόφαση από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο ε, και ήδη συζητάμε πώς θα την παρακάμψουμε αντί να συζητήσουμε πώς θα την εφαρμόσουμε και πώς θα την σεβαστούμε. Όσον αφορά το Μαρόκο, δεν υπάρχει αμφιβολία όσον αφορά το γεγονός ότι το Μαρόκο είναι σημαντικός εταίρος μας, ε, ιδιαίτερα όσον αφορά την μετανάστευση από την Αφρική. Αυτό μας ε, ε, περιορίζει όσον αφορά την ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται και μια χώρα η οποία κατηγορείται για ε, βασανιστήρια στις φυλακές της, που μια χώρα που κατέχει ξένη, ξένα εδάφη και θα έπρεπε αυτά τα θέματα να μας απασχολήσουν περισσότερα και όχι να μας ενοχλούν εδώ πέρα και να μας ταράζουν με ανοησίες. για το πώς θα προστατευθούν οι σχέσεις μας με το Μαρόκο. Υπάρχουν και άλλες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο με το ίδιο βάρος και σημασία και θα ήταν πραγματικά κατά των αρχών μας να ασχολούμαστε συνέχεια με αυτή την υπόθεση. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να θέσω δύο-τρεις ερωτήσεις εάν θα υπάρξει ειδική ετικέτα για τα προϊόντα της Δυτικής Σαχάρας ανάλογα με τα αυτές που υπάρχουν για τα κατεχόμενα εδάφη της Παλαιστίνης. Τι μέτρα λαμβάνετε για να εξασφαλίσετε την ε, εφαρμογή της απόφασης και επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεκινήσει με το, με το Ποπολισάριο και, ποια, ποιο θα είναι το μέλλον του λαού των Σαχαράουι και κυρίως ε, όσον αφορά τις μελλοντικές μας εμπορικές σχέσεις με αυτή την περιοχή. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να, να, να εκφράσω την έκπληξή μου, για να μην πω και τίποτα χειρότερο, για το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε καν τέτοια αναθεώρηση. Και δεν έχει ακόμα λάβει υπόψη 100% τη συνέπειε τη δικαστική απόφαση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα διατηνόμαστε ότι προασπιζόμαστε ε, υψηλού ανώτερου σκοπού. Και τι γίνεται εδώ επικρατεί το εμπόριο κατά των ε, ευρωπαϊκών, κατά ανθρωπινών δικαιωμάτων. Τι γίνεται λοιπόν με τα άτομα αυτά που είναι στι φυλακές. Δεν θέλω να τα επαναλάβω, είναι φρικτέ οι καταστάσει και ότι εδώ βάζουμε σε πρώτη θέση τις εμπορικές σχέσεις αποτελεί πραγματικά γεγονός ακατανόητο για μένα. Ευχαριστώ. Mr. Kawa, one last chance. Thank you, Mr. Brock. Sorry. Ο κύριος Κάβερ, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Μπρόκ. Ο κύριος Κάβερ. Να μας πείτε τη γνώμη σας θα ήθελα για, για μια γραπτή ερώτηση που έχω θέσει για τη Σομαλιλάνδη και την αναγνώριση τη, για την αναγνώριση τη Παλαιστίνης την οποία έθεσα πριν από δύο χρόνια. Αυτό επηρεάζει τι πολιτικέ αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και θεωρώ ότι αποτελεί αντίφαση. Πείτε μα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση πώ μπορεί να εφαρμόσει άλλα μέτρα και σταθμά για την Παλαιστίνη, τη Σομαλιλάνδη και τώρα άλλα για τη Δυτική Σαχάρα. Monsieur Président. Moi, voudrais euh, euh, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να θέσω το εξή ερώτημα. Όταν έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θέτει προβλήματα πολλέ φορέ στη συνεργασία με το Μαρόκο, να για μια φορά που τα πράγματα λειτουργούν. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί με θέλουν να το ανατρέψουμε. Για μένα το θέμα του, της δικής Σαχάρας είναι θέμα του Ενωμένου Εθνών. Δεν πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μαρόκο είναι ένας πολύ σημαντικός και βασικός αξιόπιστος εταίρος για μας. Έχουμε 18 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια εξαγωγών για το Μαρόκο. Έχουμε αξιοπιστία στην ε, ρύθμιση των ε, προσφυγικών ροών που μας προστατεύει από το Μαρόκο και εναντίον τη τρομοκρατία, Γιατί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφήνει αυτό το θέμα που είναι θέμα των Ηνωμένων Εθνών στα Ηνωμένα Έθνη. Και θέλω να υπενθυμίσω τους συναδέλφους μου ότι υπάρχει και δυσφορία των ε, λαών μας πολλές φορές για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Υπάρχουν παρόλα αυτά κάποια πράγματα τα οποία λειτουργούν σωστά, όπω είναι η συνεργασία μα με το Μαρόκο, δεν πρέπει να την υποσκάψουμε. Υπήρξε μια συμφωνία, λέει ο πρόεδρο Ευρωπαϊκή Ένωση Μαρόκο. Και αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό δεν είναι μια παρέμβαση ή ανάμιξη, είναι διατήρηση του κράτους δικαίου. Δεν πρέπει να το θεωρείτε ότι είναι μια παρέμβαση είναι μια συμφωνία με το Μαρόκο στην οποία είναι αρμόδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το αν είναι σωστή η λαθασμένη συμφωνία αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Σημαντικό είναι το ότι πρέπει να διατηρήσουμε το κράτος δικαίου. Δεν ξέρω αν και στο δικό σας κόμμα είναι κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό το κράτος δικαίου. Δάτη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Σωστά υπενθυμίζετε τις αρχές της, ε, του δικαίου για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως αυτό πρέπει να πω ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υπενθυμίζει ακριβώς την ανάγκη να διατηρηθεί το κράτος δικαίου. Τόνισε λοιπόν ότι με την ανατροπή της απόφασης του Πρωτοδικίου ότι εξακολουθεί να ισχύει η εμπορική συμφωνία του 2012 μεταξύ Ευρωπαϊκής και Μαρόκου και δεύτερον υπενθυμίζει ότι για να παρέμβει κανείς ενώπιον του δικαστηρίου θα πρέπει να έχει μια νομική αναγνώριση και ένα ένομο δικαίωμα, κάτι το οποίο δεν ισχύει για το Πολυσάριο. Δεν μπορεί λοιπόν να υποστηρίζονται αποφάσει οι οποίες είναι πολιτικού χαρακτήρα και απόλυτα μεροληπτικές, όπως έγινε στο, ε, στην περίπτωση αυτή. Το Μαρόκο δεν είναι ένας τυχαίος σύμμαχός μας, είναι ένα σημαντικός ε, σύμμαχος στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, στην διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών και πάρα πολύ σημαντικός παράγων για τη συνεργασία μας με την ε, Αφρική. Είναι παράδειγμα προς μίμηση το Μαρόκο σε ό,τι αφορά τους αφρικανικούς λαούς και με τον τρόπο αυτό, με την απόφαση αυτή μπορούμε να ενισχύσουμε και πάλι τη σχέση εμπιστοσύνη που έχουμε που εμείς οι ίδιοι θέσαμε εν ε, Κύριε Westcott, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τη σημασία της ασφάλειας της Ευρώπης και της ανάπτυξης της Αφρικής που παίζει σημαντικό ρόλο το Μαρόκο σε αυτό. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα εφαρμοστεί πλήρως, η, αν θα περατωθούν διαπραγματεύσεις και θα ε, εφαρμοστεί πλήρως η Συμφωνία Ελευθερού Εμπορίου με το Μαρόκο μετά από τόσα χρόνια διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ, Πέτρα, και καλή χρονιά σας εύχομαι και σε εσάς και σε όλους τους συναδέλφους. Να ευχαριστήσω τους κυρίους που μας ε, μίλησαν για την ε, σημερινή κατάσταση, τον κύριο που μας μίλησε για τη σημερινή κατάσταση. Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα για τη σημασία του Μαρόκο και γιατί θα πρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω τη σχέση μας με τη χώρα αυτή. Νομίζω ότι το πραγματικό θέμα είναι η Βυτική Σαχάρα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Να πω μάλλον ότι όλοι θα πρέπει να εργαστούμε για να πετύχουμε την ειρήνη. Που τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να βοηθήσουμε το Μαρόκο να λύσει το θέμα της Δυτικής χαράς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ χαίρομαι για το γεγονό ότι η Συμφωνία για τα Αγροτικά Θέματα μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μαρόκου εξακολουθεί να ισχύει μετά από την ανατροπή τη απόφαση του Πρωτοδικείου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από την προσφυγή του Συμβουλίου. Θέλω να πω το εξή όμω. Είναι πάρα πολύ σημαντική η Συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με το Μαρόκο. Θα πρέπει να την προσέξουμε πολύ. Είναι ένα προνομιακό εταίρο το Μαρόκο. Το θέμα της Δυτικής Σαχάρας θα πρέπει να επιληθεί μέσω διμερών συνομιλιών μεταξύ του Μαρόκου και του Πολυσάριου υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών βάσει των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν θα πρέπει να έχουμε παρεμβάσεις στις διμερείς σχέσεις Μαρόκου-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια σημαντική χώρα που είναι γείτονα και φίλο μας. Η συμφωνία μας έχει πάρα πολύ σημαντικό εμπορικό, ε, οικονομικό και ανθρώπινο χαρακτήρα και επίσης έχει να κάνει και με την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και των μεταναστευτικών ρόμων. Θέλω να σας πεθυμίσω ότι η Αραβική Άνοιξη μας οδήγησε σε μεγάλες απογοητεύσεις από πολλές χώρες που βρίσκονται στην περιοχή αυτή, αλλά το Μάροκο παρέμεινε φάρος σταθερότητας, μια χώρα γαλήνια που προέβη σε θετικές μεταρρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διατηρήσει και να συμβάλλει σε αυτήν την σταθερότητα. Όπω ξέρετε κύριε Westcott, η απόφαση αυτή οδήγησε σε σημαντικέ διαταραχέ στη σχέση του Μαρόκου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να υπενθυμίσω στον ε, εκπρόσωπο της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ότι εφόσον ξεπεράσαμε αυτό το σκόπελο θα πρέπει να επαναλάβουμε τις προσπάθειες να βελτιώσουμε τη σχέση μας στο καλύτερο επίπεδο όπως θέλει η πλειοψηφία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ συμφωνώ λέει η κυρία Χιμένα. Συμφωνώ ότι οι σχέσεις μας με το Μαρόκο είναι πολύ σημαντικές. Και ιδίω για μια χώρα όπως η Ισπανία που είναι άμεσος γείτονας του Μαρόκου. Το Μαρόκο αυτή τη στιγμή <clears throat> είναι μια ανισίδα σταθερότητος και ισορροπίας και πρέπει να την προασπίσουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι η χώρα αυτή έχει εισβάλλει σε ένα έδαφος που δεν της ανήκει και όταν λένε οι συνάδελφοι γιατί, δεν, γιατί θίγουμε πράγματα τα οποία λειτουργούν, όχι λειτουργούν για μέρους αλλά όχι για άλλους, για τους Σαχαραούι παραγματος χάρη. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να διατηρήσουμε τη σχέση μας με το Μαρόκο, αλλά συγχρόνως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται πόροι που δεν ανήκουν στο βασίλειο του Μαρόκο. Επομένως το ερώτημα είναι το εξή. Πρέπει να διατηρήσουμε τη συνεργασία με το Μαρόκο, αλλά διατηρώντας τους πόρους που ανήκουν στους Σαχαραούι στην δικαιοδοσία των Σαχαραούι. Να εξασφαλίσουμε το Μαρόκο δεν χρησιμοποιεί πόρους οι οποίοι δεν ανήκουν σε αυτό, αλλά στους γείτονές του. Αν μπορέσουμε να το επιτύχουμε αυτό, θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ενέργεια από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ με ιδιαίτερα από ορισμένε παρεμβάσεις που αναφέρθηκαν, γιατί η απόφαση αυτή είναι πάρα πολύ σαφής. Η απόφαση κάνει σαφέ ότι η Δυτική Σαχάρα δεν είναι τμήμα του Μαρόκου. Και δεύτερον ότι καμία συμφωνία, είτε εμπορική, είτε ε, για τα αλληλευτικά θέματα, μπορεί να εφαρμοστεί στο έδαφος της Δυτικής Σαχάρας. Και επίσης δεν μπορεί να υπάρξει καμία ενέργεια στη Δυτική Σαχάρα χωρίς την πρώτερη απόφαση και συνένεση του λαού της Δυτικής Σαχάρας. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω κύριε Westcott ποια είναι η άποψη της Κομισιόν και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για πώς θέλετε να εφαρμόσετε αυτή την ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και δεύτερον θα ήθελα να ξέρω πότε θα υπάρξει επαφή μεταξύ ημών με ύψιλον και του μετόπου Πολυσάριου. Τρίτον, θα ήθελα να ξέρω πότε θα τροποποιήσετε την, τον κατάλογο των εξαγωγέων που είναι εγκεκριμένοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην λειτουργούν από τη Δυτική Σαχάρα. Και θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με τις ισπανικές επιχειρήσεις, οι γερμανικές επιχειρήσεις που εργάζονται στην Δυτική Σαχάρα. Τι θα κάνετε για να εξασφαλίσετε ότι αυτέ οι επιχειρήσει θα σταματήσουν τι δραστηριότητε του εκεί, γιατί αυτό πια είναι παράνομο. Και να σα υπενθυμίσω κάτι ακόμα. Έχουμε ένα πλοίο που λέγεται Key διακόπτει ο πρόεδρο στον ομιλητή. Σα ευχαριστώ κύριο Σουέσκο και θέλω να ευχαριστήσω όλου του συναδελφού για τι ε, παρεμβάσει του. Υπάρχουν τρία στοιχεία στα οποία θέλω να απαντήσω η εταιρική μας σχέση με το Μαρόκο, η οποία είναι σημαντική και πάρα πολύ σταθερή. Δεύτερον, όπως είπε ο πρόεδρος, είμαστε μια κοινότης δικαίου και γι' αυτό θα πρέπει να σεβαστούμε οποιαδήποτε απόφαση η οποία λήφθη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να εξασφαλίσουμε τη σωστή εφαρμογή του. Τρίτον, υπάρχει το θέμα της ειδικής Σαχάρα. Α τα διεξέλθω διαδοχικά τα θέματα αυτά. Αναγνωρίζουμε απόλυτα την κρίσιμη σημασία της σχέσης μας με το Μαρόκο σε τομείς όπως είναι η μετανάστευση, όπως είναι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, όπως είναι το εμπόριο. Όλα αυτά είναι τομείς όπου έχουμε μια σημαντική και βαθιά σχέση με το Μαρόκο και είναι η πρόθεσή μας, όπως είπα, να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο αυτήν την σχέση. Συνεχίζουμε λοιπόν τις συζητήσεις με το Μαρόκο, τώρα που μπορούμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου και για άλλους τομείς όπου μπορούμε να διευρύνουμε την εταιρική σχέση για την κινητικότητα, να βρούμε τρόπους να υποστηρίξουμε τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση των διαφόρων ηθαγενών κοινοτήτων. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα που είχαν ανασταλεί η εξέτασή τους μπορούμε λοιπόν να τα προωθήσουμε ώστε οι σχέσεις μας να παραμείνουν θετικές, φιλικές και παραγωγικές. Δεύτερον, όπως είπα και πριν, οποιαδήποτε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι δεσμευτική για τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι μια μακρά και πολύπλοκη απόφαση. Όσοι την διάβασαν θα ξέρουν ότι υπάρχουν πολύ λεπτομεριακά τα νομικά επιχειρήματα που αναφέρονται και πρέπει να δούμε ποιες είναι και οι συνέπειες αυτών των ε, επιχειρημάτων και ποιος είναι ο άμεσος αντικτυπός Ο άμεσος αντικτυπός καταρχήν είναι ότι έχει ανατραπεί η απόφαση η οποία ακύρωνε ένα τμήμα της απόφασης Συμβουλίου. Η απόφαση Συμβουλίου παραμένει ενισχύη. Αλλά θα πρέπει να δούμε πλήρως και σε βάθος ποιος θα είναι ο αντίκτυπος των επιχειρημάτων που ανέφερε το δικαστήριο για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Να δούμε αν υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις. Όταν, δούμε, όταν λοιπόν θέλουμε να δούμε πώς θα επηρεαστούν οι λιμένες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ενημερώσουμε πλήρως το Κοινοβούλιο. Και δεν είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της μόνο, αλλά εμπλέκει και το Μαρόκο με το οποίο εμεί συνάψαμε αυτή τη συμφωνία καταρχήν. Πρέπει να συμφωνήσουμε μαζί τους για το ποιε είναι οι ε, συνέπειες και πώς πρέπει να αντιμετωπιστούμε. Το τρίτο σημείο για τη είναι ένα έδαφος για το οποίο υπάρχει διεθνής διαμάχη. Και η θέση μας είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να επιλύσουν τα Ηνωμένα Έθνη. Και αυτό υπογραμμίζει και τη σημασία της επίλυσης αυτού του προβλήματος, ώστε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξουμε τις ανανεωμένες προσπάθειες των ΗΠΑ για να βρούμε μια λύση για αυτή τη διαμάχη και θα υποστηρίξουμε το νέο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ για να επιτύχει μια δίκαια και αμοιβαία ε, αποδεκτή λύση για να υπάρξει αυτοδιάθεση του λαού της Δυτικής Σαχάρας μέσα στα πλαίσια ε, ρυθμίσεων που θα συνάδουν με τη Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών. Και βέβαια όταν μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτό με τον νέο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών θα είναι από τις υψηλότερες μας προτεραιότητες. Θα θέλουμε να ακούσουμε τις δικές τους απόψεις για το πώς θέλει να προωθήσει το θέμα αυτό και να, θα δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να τον υποστηρίξουμε. Σας ευχαριστώ και νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να διακρίνουμε αυτά τα δύο κομμάτια. Έχουμε τη συμφωνία η οποία έχει επικυρωθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για συγκεκριμένα θέματα δεν έχει συμφωνήσει η δικαστική απόφαση και τώρα περιμένουμε μια πρόταση για το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εκτορικής Δράσης θα εξαγάγουν τα απαραίτητα συμπεράσματα σε ό,τι αφορά και τις Διαπραγματεύσει προκειμένου να εφαρμοστεί η δικαστική απόφαση. Το δεύτερο θέμα είναι η πολιτική για τη Δυτική Σαχάρα. Και εκεί θα πρέπει πραγματικά να υποστηρίξουμε τη διαδικασία ε, των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να υπάρχει κάποια επιτάχυνση. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που ήρθατε εδώ κύριε Ρεσκότ.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 Κυρίε και κύριοι, στο σημείο 6 τώρα. Έκταση για τη Σερβία. Να παρακαλέσω όμω καταρχά, η κυρία Αγγελικά Άχιαος, ε, ε, διευθύντρια τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση υπεύθυνη για θέματα Δυτικών Βαλκανίων ε, και Τουρκία, να μα μιλήσει για την σύλληψη του Ράμος Αρντινάη και να κάνει τις ε, σχετικές δηλώσεις που σκοπεύει να κάνει. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που είστε εδώ πέρα και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλή χρονιά και σε όλους σας. Να ευχαριστήσω επίσης και τα μέλη του Κοινοβουλίου, τους βουλευτές που μου έδωσαν την ευκαιρία να πάρω το λόγο. Εν συντομία, θα ήθελα καταρχάς να μιλήσω και για τους δύο εκθέσεις, η κυρία Ρονατσοκ και ο κύριος Μακάλιστερ, ε, πρέπει να πω ότι κάναν τεράστιες προσπάθειες. Έχουν κάνει τεράστιες προσπάθειες προκειμένου και η Σερβία και το Κωσυποπέδιο να κινηθούν προς την ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Και σε ό,τι αφορά την κατάρτιση των εκθέσεων αυτών, βλέπουμε ότι πραγματικά έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια και από τις δύο πλευρές. Και εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε ότι και από τις δύο πλευρές έχει σημειωθεί σημαντικό το 2016 σε ό,τι αφορά τον δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη Σερβία και για το κοσικό Η Σερβία ξεκίνησε και το κεφάλαια, έκλεισε και προσωρινά ένα κεφάλαιο. Το κοσυφοπαίδιο με την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Σταθεροποίησης έγινε το πρώτο Συμβούλιο SAA τον Νοέμβριο και η Συμφωνία Πλαίσιο με το Κωσυφοπέτη υπογράφτηκε για πρόσβαση στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ε, παραδείγματα είναι αυτά και μόνο για το πώς συνεργαζόμαστε, αλλά φυσικά να σας πω που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά το διάλογο και τι έγινε προσφάτως σε ό,τι αφορά και την σύλληψη του πρώην Πρωθυπουργού Ράμος Χαραντινάη. Σε ό,τι αφορά το θέμα του διαλόγου, να σας πω ότι έχουν σημειωθεί πολύ καλές εξελίξεις από τον Αύγουστο του περσινού έτους και για τις δύο χώρες. Καταφέραμε να προχωρήσουμε, να πετύχουμε συμφωνία για, τη της Μητρόμητρα και τις τηλεπικοινωνίες, το ε, έλαβε ένα ITU, ένα διεθνή κώδικο, η Σερβία δε. Έχει και μια εταιρεία πιστοποιημένη στο πεδίο και σε ό,τι αφορά θέματα Να σας πούμε ότι όλες οι πλευρές συμφώνησαν ότι όλα τα βήματα που έχουν γίνει για την πρόοδο, για τη συνεργασία, για την ανταλλαγή πληροφοριών, ε, μεταφορά τέτοιων διαδικασιών ή οι διαδικασίε αυτέ ήταν πραγματικά ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τα εμπρό. Και αυτό είχαμε προβλέψει και από τις δύο πλευρές ε, σε ό,τι αφορά το διάλογο που διευκολύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε φυσικά και την ε, σύλληψη του πρώην Πρωθυπουργού Ραμού Καραντίνα ε, στις 4 Ιανουαρίου στη Γαλλία. Αυτό προφανώς προκάλεσε μια σειρά έντονων αντιδράσεων στο κοσυφοπαίδιο. Και εδώ και στο εξωτερικό και παντού. Και αυτό μας καταδεικνύει για άλλη μια φορά γιατί θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών και γιατί είναι απόλυτη προτεραιότητα να συμμετάσχουν και οι δύο πλευρές στο διάλογο. Φυσικά, παρακολουθούμε τις εξελίξεις ε, σε ό,τι αφορά τη σύλληψη και το, τη διαδικασία την ακολουθούν οι γαλλικές αρχές όλα τα μέσα, όλες οι πλευρές θα πρέπει να παραμείνουν ψύχρεμες και να συνεργαστούν σε ένα επικοδομητικό κλίμα για την εξομάλυνση των σχέσεων. Γιατί προφανώς τέτοιες υποθέσεις δεν βοηθούν την επικοδομητική ατμόσφαιρα συνεργασίας. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και τους βουλευτές εδώ που έχουν ε, καταβάλει προσπάθειες για να υπάρχει πιο πολύ διάλογος και πιο σωστός διάλογος και προκειμένου και οι δύο πλευρές να συνεχίσουν να επικοινωνούν και να εξηγούν τι κάνουν, γιατί το κάνουν και γιατί αυτό είναι επωφελές. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Έρχομαι τώρα στην έκθεση αυτή, την ιδία. Ο κύριος Μακάλιστερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι τιμή μου να παρουσιάζω την, ε, την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, Σερβία. Έχουμε ε, σελίδε, προσπάθησα να μου γίνεται πιο σύντομο και συγκεκριμένε. Στι πρώτε 7 παραγράφου έχω προβεί σε μια γενική εκτίμηση τη πορεία τη Σερβία προ την Ένωση, ε, αναφερόμενο στα έξι κεφάλαια που έχουν μέχρι στιγμή ανοίξει και σχετίζονται με την οικονομική πολιτική τη ε, ε Σερβία, την ευθυγράμμιση τη με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και το κρίση της μεταναστευτική. Μετά αναφέρομαι στα κριτήρια της Κοπενχάγης, κράτος δικαίου, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και σεβασμός για την προστασία των μειονοτήτων. Τέλος, έχω προσθέσει την περιφερειακή συνεργασία και την ενέργεια. Ε, θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να τονίσω κάποια σημεία που είναι μεγάλη σημασία όσον αφορά την πορεία της Ένωσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς, κράτος δικαίου. Θέλω να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία ε, για να δούμε πώς ε, και αν ε, αυτό μπορεί να, δια, να διαταράξει την ε, διαπραγματευτική διαδικασία. Η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, του δικαστικού ε, τμήματος θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη. Υπάρχει ωστόσο καθυστέρηση, ε, υπάρχει διαφθορά και οργανωμένο έγκλημα που παραμένουν διαδεδομένα και αντιπροσωπεύουν ένα εμπόδιο στη δημοκρατική αναζήτηση της, της χώρας και την οικονομική της ανάπτυξης. Δεύτερον, δημοκρατία. Καλωσορίζω το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει αυξήσει τη συμμετοχή του Σερβικού Κοινοβουλίου στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, η εκτεταμένη χρήση των επιγουσών διαδικασιών στην υιοθέτηση της νομοθεσίας παραμένει μεγάλη ανησυχία μας. Επιπλέον, θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις σερβικές αρχές να συνεχίσουν στο δρόμο της ανεξαρτητοποίησης του, το Κοινοβουλίου. Τέλο, ε, τρίτον, μάλλον θα πρέπει να υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών δικαιωμάτων, ελευθεριών μάλλον, που πρέπει τώρα να εφαρμοστεί. Συμφωνώ με την Κομισιόν και το Συμβούλιο ότι θα πρέπει να εγγυηθούμε την. Ε, ε εγγύηση της ελευθεροδιπίας καθώς και την προστασία των δημοσιογράφων. Οι απειλές εξακολουθούν και οποιαδήποτε επίθεση κατά των μίντια και των δημοσιογράφων θα πρέπει να ερευνάται. Τέταρτον, η περιφερειακή συνεργασία και οι ε, αγαστές ε, σχέσεις γυπνίασης. Η κυβέρνηση στο Βελιγράδι έχει προβεί σε σημαντικές συμβολική πρακτικά βήματα αλλά και ουσιαστικά βήματα για να συμβάλλει σε καλύτερη συνεννόηση και συνεργασία στην περιοχή. Όλοι γνωρίζουμε ότι η διαδικασία ένταξη της Σερβίας στην Ένωση βασίζεται στην ε, ομαλοποίηση των σχέσεων με το Κωσικοπαίδιο και οι δύο πλευρές θα πρέπει να συνεχίσουν να κινούνται εμπρός με την πλήρη εφαρμογή όλων των συμπεφωνημένων με καλή την πίστη και έγκαιρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, μια τελευταία παρατήρηση. Ε, από όλε τι πλευρέ ε, το 2016 ήταν σημαντική χρονιά για την Σερβία. Μετά από τι κοινοβουλευτικέ εκλογέ ε, τον Απρίλιο, η νέα κυβέρνηση έχει επιβεβαιώσει τη δέσμευσή τη στη στρατηγική συνεργασία της χώρας προς την πρόσβαση. Έχει συνεχίσει σε την πορεία αυτή και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ πως είναι δικό μας καθήκον να στηρίξουμε και να θα επηρεάσουμε θετικά τη Σερβία στην πορεία της προς την Ένωση. Και τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία της Επιτροπής ΑΦΕΤ αλλά και ε, την ομάδα ε, του ΕΛΚΑ, ε, την ομάδα μου για τη στήριξή της. Ελπίζω σε καρποφόρα συνεργασία μαζί σας και κυρίως με τους Κιώδης ώστε να προχωρήσουμε σε ένα καραλό αποτέλεσμα και προσβλέπω στο να ακούσω τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, David. 8 Ιανουαρίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. 18... 28 Φεβρουαρίου θα γίνει η ψηφοφορία. Και είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται στην κούρσα, αν θέλετε, των Δυτικών Βαλκανίων για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ εμπλέκεται και το άρθρο αυτό που έχει να κάνει με την ένταξη μιας χώρας και επομένως εδώ η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πάρα πολύ σημαντικά μια χώρα λοιπόν η οποία έχει τη φιλοδοξία να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να έχει μια αυταρχική συμπεριφορά του λαού του, της θα πρέπει να εξασφαλίσει μια ε, βελτίωση σε όλους αυτούς τους τομείς που έχουν να κάνουν με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Έχουμε πολλούς οι οποίοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Κούκαν είναι ο πρώτος ο οποίος λαμβάνει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον εισηγητή για μια αντικειμενική και ισορροπημένη έκθεση που εστιάζει στις κύριες επιτάξεις Σερβίας μέχρι τώρα και σε αυτά που παραμένουν να επιτευχθούν. Πριν προμπούμε στην συζήτηση για τη Σερβία, θα ήθελα να κάνω μια γενικικότερη έκκληση σε όλους από εμά που παρακολουθούμε τη διαδικασία της διεύνησης. Εφέτος έχουμε μια δυνατότητα να προχωρήσουμε με πολλές χώρες της περιοχής, των Βαλκανίων θα πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτό το ευρύτερο ευρωπαϊκό εγχείρημα που θα ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη Σερβία την ίδια έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο το 2016, άνοιξαν κεφάλαια διαπραγματεύσεων και έχει ευθυγραμμιστεί περισσότερο με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί και το 2017. Θα πρέπει να την υποστηρίξουμε σε αυτή τη διαδικασία, ιδίω σε ό,τι αφορά τις ενεξελίξεις μεταρρυθμίσεις. Ελπίζω ότι αυτή η διαδικασία θα αντιμετωπιστεί βάσει της επιτυχίας της και δεν θα ξαναγίνει το επόμενο θύμα διμερών πολιτικών αντιμαχιών. Η Σερβία έχει επιτύχει σημαντικές βελτιώσει στα οικονομικά θέματα, έχει αντιμετωπίσει με πραγματιστικό τρόπο την κρίση μετανάστευση. Η Σερβία έχει καταφέρει επίση να είναι καλό γείτονα με επικοδομητική αντιμετώπιση για τα διμερή θέματα. Θέλουμε λοιπόν να ενθαρρύνουμε τη Σερβία να εργάζεται για τι καλύτερε σχέσει με του γείτονέ τη και να διατηρήσει τη διαδικασία ομαλοποίηση με το κοσφοπέδιο, καλή την πίστη και να εφαρμοστούν οι συμφωνίε που έχουν επιτευχθεί. Αλλά ακόμα πρέπει η Σερβία να κάνει περισσότερα πράγματα, ιδίω για το κράτο δικαίου, τον αγώνα κατά τη διαφθορά και την βελτίωση τη δικαστική ανεξαρτησία, Θα είναι από τι μεγαλύτερε προκλήσει μέσα στη διαδικασία διαπραγματεύσεων για την ένταξή τη. Θέλουμε να δούμε μια διαδικασία μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό και Δικαστήριο ήδη αναφέρεται για πολύ γερό σε προβλήματα που έχουν να κάνουν με κατάχρηση εξουσίας που εκκρεμούν στα πυρικά δικαστήρια και θέλουμε να σταματήσουν να γίνονται χρήσεις τέτοιων επιχειρημάτων για καταδίκη στα δικαστήρια. Επίσης, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα του εμπορικού καθεστώτος της Σερβίας με την Ευρωασιατική Ένωση και θέλουμε επίσης να ξεκινήσει μια κριτική διαδικασία για την βελτίωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και γενικά της ελευθερίας έκφρασης. Εγώ θα καταθέσω τις αντίστοιχες τροπολογίες για τα σχόλια αυτά και πάλι όμως θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή για την πολύ καλή εργασία που έχει φέρει σε πέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κούκαν. Η κυρία Φαγιόν που είναι σκιώδης εισηγήτρια έχει τον λόγο από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Μακάλιστερ για την ε, πολύ ισορροπημένη έκθεση για τη Σερβία και θα ήθελα να τονίσω κάποια από τα γεγονότα και τις εξελίξεις που μας ανησυχούν. Όσο και να καλωσορίζω το άνοιγμα επιπλέον κεφαλαίων στι διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να σα πω ότι λυπούμε ιδιαίτερω για το γεγονό ότι αυτό το επισκίασε το άνοιγμα της, ε, του κεφαλαίου 27 και ελπίζω, σε ό,τι αφορά την Κροατία, ελπίζω λοιπόν να υπάρξει λιγότερη ένταση στις σχέσεις Σερβίας-Κροατίας φέτος. Σε ό,τι αφορά τις αιτιάσεις ε, από τον Πρωθυπουργό προς τον διαμεσολαβητή, θεωρώ ότι είναι κάτι επιζήμιο για τη δημοκρατία και θίγεται ο κύριος διαμεσολαβητή. Και γι' αυτό καλωσορίζω λοιπόν την παραγραφό 14 που αφιερώνεται στη σημασία του ρόλου του διαμεσολάβητη στην Σερβία και σε κάθε δημοκρατία. Πέρα από τις ε, πρόοδες που έχουν σημειωθεί στο θέμα του κράτους δικαίου, πολλά θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω. Αυτά που έγιναν στο Βελιγράδι την ημέρα των εκλογών, το βράδυ των εκλογών στην περιοχή του Σεμβάλα και αυτό το, το γεγονός ότι δεν έχουν επιληθεί τα θέματα αυτά ακόμα, είναι απαράδεκτο παρά την ε, παρουσία της κοινωνίας των πολιτών και δημοσίων λειτουργών. Θεωρούμε ότι αυτό δεν έχει λήξει ακόμα και φυσικά βαραίνει την κοινωνία η ελευθερία των μέσων ενημέρωση τη έκφραση. Αναφέρθηκαν τα θέματα αυτά και ξέρουμε όλοι ότι επιδεινώνονται τα πράγματα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά στην Σερβία, σε ό,τι αφορά τον δημόσιο κλάδο τη ΜΚΟ. Έχουμε λάβει ε, άπειρες καταγγελίες σε ό,τι αφορά την καταπίεση που επικρατεί σε ό,τι αφορά την δυνατότητα εργασία των δημοσιογράφων κτλ. Και τέλο, θα ήθελα να επενέσω τι προσπάθειε τη Σερβία σε ό,τι αφορά την επικοδομητική προσπάθεια, σε ό,τι αφορά την περιφερειακή συνεργασία. Θα πρέπει να σταματήσει η μαζική εκροή εγκεφάλων, ειδικά νέων από τη Σερβία και υπάρχει μια σχετική πρωτοβουλία, για παράδειγμα, η οποία αποτρέπει όλα αυτά τα φαινόμενα. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν γρήγορα σχετικέ αποφάσει στην επόμενη περίοδο και θα σα διαβεβαιώσω ότι και εγώ θα βοηθήσω όσο περνάει από το χέρι μου μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και να ακούσουμε του συζητητέ, ο κύριο Τάνοκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω και να συγχαρώ και να ευχηθώ και καλή χρονιά στον συνάδελφο David McAllister. Είναι ισορροπημένη η έκθεση και περιλαμβάνει πολλά θέματα και συνοψίζει πολύ σωστά το που βρισκόμαστε στη διαδικασία ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά η ομάδα μα υποστηρίζει την προσχώρηση της, Ευρω... της Σερβίας και των υπόλοιπων Δυτικών Βαλκανίων και καλωσορίζουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη Σερβία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την οικονομία, τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες όπως το Μαυροβούνιο και θα υποβάλω σχετική έκθεση ε, εν ευθετό χρόνο και ότι κάνει κάποια βήματα σε ό,τι αφορά την Αλβανία και το Κωσυφοπέδιο. Φυσικά με ανησυχεί ε, η πρόσφατη σύλληψη πρώην αξιωματούχου του Κωσυφοπεδίου και ελπίζω αυτό να μην είναι μεγάλο πλήγμα για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά πολλά ε, συνενησυχίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην περιοχή στη Σερβία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ελευθερία έκφραση, στα δικαιώματα των μειονοτήτων, μεταξύ άλλων και των ΛΟΑΔ. Και φυσικά η Σερβία, για να είμαστε δίκαιοι, αντιμετώπισε τεράστιες προκλήσεις πρόσφατα με την προσφυγική κρίση. Άρα, αλλά, αλλά για να είμαστε και πάλι αρκετά ακριβείς, ε, είναι χώρα διαμετακόμισης στη Σερβία. Δεν ζήτησαν και πολλοί να παραμείνουν στην Σερβία. Η Σερβία λοιπόν όπως και άλλες υποψηφίες χώρες θα πρέπει να συνεχίσει δυναμικά τις μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση, την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος της διαφθοράς και αυτό που εμάς μας απασχολεί ιδιαίτερα στην ομάδα μου είναι η αποτυχία συμμετοχής στην ΚΕΠΑ της ε, Σερβίας και στο καθεστώς κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ε, και αυτό νομίζω καταδεικνύει τη σφαίρα επιρροή του Πούτιν και αυτό μας απασχολεί βεβαίως. Και αποσταθεροποιεί, θεωρώ, και την γεωπολιτική κατάσταση όλων των Δυτικών Βαλκανίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, ο κύριος Φάκλ. Θα ήθελα εγώ να συμφωνήσω με τους συναδέλφους που πένεσαν την προσέγγιση του εισηγητή μας, του κυρίου Μακάλιστερ, ο οποίος ε, έθεσε το τόνο για αυτή τη συζήτηση, αντικειμενικός. Εγώ πιστεύω πως η Σερβία το χρειάζεται αυτό και είναι πολύ σημαντικό για τις σχέσεις ανάμεσα στη Σερβία και στην Ένωση πρέπει να διατηρηθεί αυτός ο θετικός τόνος στη συζήτηση. Τώρα υπάρχουν κάποιες επαναλαμβανόμενες πληροφορίες σε αυτή την έκθεση. Για παράδειγμα, καθυστερήσεις όσον αφορά την εφαρμογή της εθνικής ε, στρατηγικής κατά της ε, διαφθοράς, καθώς και ε, προβλήματα στην διεξαγωγή των ερευνών, στις ποινικέ διαδικασίες και ούτω καθεξής, καθώς επίσης δεν αναφέρονται οι ποινικέ δράσεις όσον αφορά ε, την ανάμειξη ψηλά ιστάμενων προσώπων. Ε, ε, θα έπρεπε να επαναλάβουμε την ανεξαρτησία της Βοηβοντίνας και την προστασία των μέσων μαζική ενημέρωσης, δηλαδή πράγματα που έρχονται και πανέρχονται. Θέλω να πω δύο λόγια όσον αφορά τη συνυπευθυνότητα τη Σερβία με άλλες χώρες στην ε, περιοχή. Έχει δημιουργηθεί πρόσφατα μια ατμόσφαιρα η οποία θυμίζει κρίσιμες περιόδους που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε στην ιστορία μας. Για παράδειγμα, αυτή η ε, διαμάχη ε, ε, ανάμεσα στην Κροατία και τη Σερβία, το μπλοκάρισμα, ε, γιατί οι Κροάτες σε πολιτική έχουν πει ότι δεν θα ξανακάνουν τα ίδια λάθη που έκαναν οι Σλοβαίνοι όταν οι Κροάτες προσπαθούσαν να μπουν στην Ένωση, αλλά τώρα φαίνεται να κάνουν κάτι πολύ χειρότερο. Για τη Βοσνία και Ερσεγοβίνη λοιπόν να πούμε ότι η Σερβία έχει ε, απαράδεκτες σχέσεις για παράδειγμα, ο Σέρβος Πρόεδρος συμμετέχει σε, μια πολύ επίμαχη, σε έναν επίμαχο ερωτισμό στη Βάνια Λόκα, όπου ο Πρωθυπουργό δεν παρέστηκε για πολύ βάσιμους λόγους. Η Σερβία είχε σύγκρουση και με τη Μακεδονία Ο Πρωθυπουργό Ντάτιτ ε, είπε ότι θα αναγνώριζε ε, τη Μακεδονία ίσως ε, με το ιστορικό της όνομα, πράγματα τα οποία δεν στέκουν και αυτού του είδους ο λόγο, αυτή η ρητορική απηχείται σε ολόκληρη την περιοχή. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πραγματικά αυτά τα ζητήματα, γιατί σε κάποια χρονική στιγμή θα πρέπει να σταματήσουν αυτές αυτά τα προβλήματα. Και έπειτα, για το καθεστώ του Κωσυφοπεδίου στην UNESCO και εδώ θα ήταν πολύ πιο παραγωγικό αν η Σερβία και το Κωσυφοπέδιο ε, έφταναν σε κάποια συμφωνία για την ε, κοινή προστασία αυτών των ε, καταπληκτικών μνημείων της ιστορίας της Σερβίας και αν τα καταστούσαν προσιτά σε ολόκληρο τον κόσμο αντί να παίζουν πολιτικά παιχνίδια με για αυτά τα μνημεία. Θα τελειώσω λοιπόν λέγοντας ότι αυτή η έκθεση είναι θετική, μπορώ να την στηρίξω και θα ήθελα επίσης να επενέσω την Σερβία για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει στην πορεία της προς την Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριος Πέτερλε. Θα μιλήσω και πιο μετά για το 25ο συζήτρια, αλλά να σας πω ότι εκπροσωπώ και τον σκισκιώδη τον κύριο, τον κύριο για τους πρασίνους για το θέμα της Σερβίας, τον κύριο Σόλτες και ε, λυπάμαι που σας πήρα το λόγο, απλά ακολουθούμε το σύστημα των πολιτικών ομάδων. Ευχαριστήσω λοιπόν τον Τέβιτ Μακάλιστα για την πολύ καλή αυτή έκθεση, η οποία πραγματικά καλύπτει στις 7 σελίδες που σε πολλές περιπτώσεις δεν φτάνουν καν, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά πολύ συνοπτικά καλύπτει όλα τα κύρια ζητήματα τα οποία ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μας απασχολούν σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με τη Σερβία. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια επισημαίνεται και όλες τις φοιτικές εξελίξεις και σύμφωνα με όλα όσα αναφέρει ο κ. Μακάλιστερ να πω και μερικά θετικά στοιχεία τα οποία δεν έχουν αναφερθεί ακόμα αλλά και κάποιες, κάποια επικριτικά στοιχεία. Επειδή είμαι από την Αυστρία, πρέπει να σας πω ότι όχι μόνο ως Αυστριακή, αλλά και ως Ευρωπαία, ε, εκτιμώ ιδιαίτερα το πώς συνεργάστηκε η Σερβία στο θέμα των προσφύγων που πέρασαν μέσα από την Ευρώπη των Βαλκανίων σε ό,τι αφορά τη Γερμανία, την Αυστρία κτλ. Όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν μπροστά εμάς ε, έκαναν πραγματικά πολύ σημαντικές προσπάθειες για καταλήμματα, για ανθρωπιστική βοήθεια και μακάρι όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είχαν καταβάλει τόσο μεγάλες προσπάθειες. Και επίσης εκτιμώ το γεγονός ότι η Σερβία συμμετέχει σε πολλές ε, διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές. Επίσης, σημειώθηκαν ε, εξελιξίες στατικέ και σε ό,τι αφορά τη σχέση με τον διαμεσολάβητη. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα των διεθνών σχέσεων, θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό η Σερβία να ε, ευθυγραμμίσει και την πολιτική ασφαλείας της και την, πολιτική, την εξωτερική της πολιτικής με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε και ο κ. Μακάλιστερ, μεταξύ άλλων και την πολιτική της έναντι της Ρωσίας, γιατί συχνά θεωρώ ότι αποστέλνει πολύ συγκεκριμένα μηνύματα. Προς τα πού θέλετε να κινηθείτε, προς τα εμάς, προς τη Ρωσία. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ακολουθήσει πιο σαφή πολιτική σε ό,τι αφορά το διάλογο με το κόσμο πέτειο. Θα μιλήσω και μετά για το θέμα αυτό φυσικά πιο πολύ, αλλά και από τις δύο πλευρές θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνουν πιο μεγάλες προσπάθειες για να εφαρμοστούν όλες οι συμφωνίες που έχουν συζητηθεί. Το θέμα του δημοσιογράφων αναφέρθηκε και το θέμα της διαφθοράς, διάφορες υποθέσεις αναφέρθηκαν και να σας πω και το τι έγινε η μεγάλη, ε, τα μεγάλα θέματα που επικράτησαν για την, επιτροπή, για την περιοχή της ε, Σανταμάλα. Να πω και δύο λόγια για αυτά που ακούσαμε στην αρχή για την πρόσφατη συλλήψη του πρώην Πρωθυπουργού του Κώσιφο Παιδίου. Να σας πω ότι στο σημείο αυτό πραγματικά θα είναι απαραίτητο η Σερβία να μην διατηρήσει εντάλματα σύλληψη από τα μέσα της δεκαετίας της προηγούμενης. Υπήρχε εντάλμα σύλληψης Υπάρχει και ένας ιδιαίτερος νόμος για την διεθνή δικαιοδοσία που ισχύει μόνο για τις πρώην περιοχές της ε, πρώην Όλα αυτά είναι προβληματικά και θα πρέπει να σας πω ότι ένας εισαγγελέας ε, του ε, δικαστηρίου ανέφερε πρόσφατα και δήλωσε πρόσφατα ότι το θέμα αυτό είναι πολιτικό και δεν έχει σερβεί ουσιαστικά δικαιοδοσία στο εικοσυφοπέδιο. Είναι προβληματικό λοιπόν το θέμα αυτό. Θεωρώ ότι πολύ απλά δεν βοηθά επικοδομητικά την εξέλιξη της ε, υπόθεσης δεν ε, βοηθά και τις περιφερειακές σχέσεις και θεωρώ ότι σμειώνει γενικότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα κύριε Πέτερλε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό η διαδικασία διαπραγματεύσεων με τη Σερβία να συνεχιστεί. Υπήρξε πρόοδος και νομίζω ότι το αντανακλά και η έκθεση του κυρίου Μακάλιστερ. Παρουσιάζει πολύ σωστά την ε, κατάσταση η έκθεση του εισηγητή εμείς. Συγχαίρουμε 15 φορές την ε, Σερβία, ενώ μόνο δύο ή τρεις φορές την προειδοποιούμε για την ε, Βοηβοδίνα και για άλλα θέματα, αλλά δεν εκφράζουμε τη λύπη μας για ορισμένο θέμα, ορισμένα θέματα. Αυτό θα έπρεπε να υπάρχει. Παρ' όλα αυτά βλέπω θετική την έκθεση αυτή. Είμαι ικανοποιημένος και με τις ενέργειες που έχει κάνει η Σερβία για να εξασφαλίσει καλύτερη συνεργασία με τις γειτονικέ της χώρες. Ξέρει η Σερβία που είναι τα πιθανά σημεία ανάφλεξης και που είναι οι προτεραιότητες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Πίκουλα. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Μακάλιστερ για την έκθεσή του, η οποία είναι μια σωστή απεικόνηση της κατάστασης στη Σερβία και δείχνει καθαρά τι έχει επιτύχει η Σερβία. Το άνοιγμα των πρώτων κεφαλαίων είναι μόνο ένα κομμάτι των θεμάτων που διαλαμβάνει η έκθεσή του. Έχουμε όμως και κάποια σημεία που επαναλαμβάνουν τις προηγούμενες εκθέσεις που δείχνει ότι η Σερβία έχει κάποια πράγματα να κάνει, έχει δρόμο δια, τρέξει. πραγματικά η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωση, η διαφάνεια σε σχέση με τους ε, διοκτήτε των μέσων ενημέρωση, η αντιμετώπιση των μειονοτήτων και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Όλα αυτά Επίσης θα περιλάμβαναν και την υποστήριξη του, της πορείας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το διάλογο με το Κωσυφοπέδιο. Το τελευταίο θέλω να τονίσω ότι η ιδέα της περιφερειακής αρμοδιότητος των σερβικών αρχών εναντί άλλων πολιτών και η σύλληψη του Χαραντίνας δεν οδηγούν σε μεγαλύτερη ισορροπία και ειρήνη στην περιοχή. Αντίθετα, θα πρέπει η Σερβία να παίξει σημαντικότερο ρόλο για την επίλυση διμερών διαφορών, όπως παραδείγματος χάρη σε σχέση με τα θέματα των αγνοωμένων του πολέμου για το Κωσυφοπαίδιο και την επιστροφή στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να κλείσουν κάποιες πληγές του παρελθόντος και να επιτευχθεί καλύτερη συνεργασία των γειτονικών χωρών με τη Σερβία το άνοιγμα των κεφαλαίων πρέπει να θεωρηθεί ως μια θετική πίεση προς την Σερβία για να ξεκινήσει την πραγματική μεταμόρφωση της χώρας αυτής. Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε όμως ότι αυτά τα οποία λέμε θα πρέπει να τροχοπεδίσουν την ε, πρόοδο της Σερβίας. Δεν θέλουμε να έχουμε επανάληψη αυτό που είχε γίνει από τη Σλοβενία που μπλοκάρισε για ένα διάστημα την ένταξη της ε, Κροατίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι είναι μια εξορροπημένη έκθεση η έκθεση του κυρίου Μακάλιστερ και θέλω να συγχαρώ τον Ντέβιτ. Ε, η έκθεσή του <clears throat> παρουσιάζει κάποια βασικά σημεία τα οποία είναι οριοθετημένα, είναι ιεραρχημένα με βάση τις προτεραιότητες και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Πρώτα απ' όλα το θέμα της διαφθοράς. Η Σερβία έχει επιτύχει κάποια πράγματα, αλλά βρίσκεται στην 71η θέση μεταξύ 184 χωρών βάσει της έκθεσης Transparency International. Φαίνεται ότι έχει πολύ δρόμο να διατρέξει για τα θέματα αυτά. Γι' αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε να υπάρξει μια πιο θεσμή, θεσμοποιημένη μάχη κατά της διαφθοράς και ο αρμόδιος φορέας θα πρέπει να δημιουργηθεί και να γίνει λειτουργικό στο ταχύτερο δυνατό. Και πάλι δεν πρέπει να είμαστε χαλαροί για τις βασικές ελευθερίες. Η ανησυχία που έχει εκφραστεί για την ελευθερία έκφρασης και την κατάσταση των μέσων ενημέρωσης. Αυτό δεν πρέπει να το υποβαθμίσουμε. Πρέπει να επιμείνουμε η Σερβία να σεβαστεί όλες αυτές τις ε, αξίες που είναι θεμελιώδεις για τη γενική της πρόοδο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, υποστηρίζω και εγώ αυτά που είπαν οι συναδελφοί μου για την ε, έλλειψη ευθυγράμμισης της Σερβίας με την κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το φλερτ με τη Ρωσία οδηγεί σε στάσεις οι οποίες είναι αμφισβητήσιμες σε πάρα πολλά θέματα. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε την έκκληση τη Σερβία να ευθυγραμμιστεί περισσότερο. Και τέλο, η διαδικασία αυτή χρειάζεται και τη δική μα εμπλοκή και τη συμμετοχή μα και γι' αυτό εκτιμώ ιδιαίτερα το διάλογο που έχουμε αναπτύξει με τη Σερβία. Η κυρία Σούιτσα. Ναι, ευχαριστώ. ευχαριστώ. Μπράβο. Πολύ καλή δουλειά. Με πολύ αντικειμενικό τόνο. Είναι προφανές ότι η Σερβία έχει σημειώσει πρόοδο στο άνοιγμα τεσσάρων κεφαλαίων. Όπως ακούσαμε, τα κεφάλαια αυτά θα πρέπει να θεωρηθούν ως μια μετάβαση της σερβικής πολιτικής κοινής προς την Ένωση. Μιλάμε για δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, περιφερειακή συνεργασία. Κάθε ένα κράτος έχει προβλήματα αλλά και πλονεκτήματα. Νομίζω πως η δυναμική των διαπραγματεύσεων θα, θα, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πρόοδο ε, στο κράτος δικαίου αλλά και στην εξομάλυνση των σχέσεων με το Κωσυφοπαίδιο όπου αναμένουμε καλύτερη τάση και περισσότερη δουλειά από πλευρά της Σερβίας η οποία πρέπει να τηρήσει όλα, όλες τις υποσχέσεις, όλες τις ε, συμβάσεις και να στηρίξει την εργασία των ανεξαρτήτων σωμάτων. Επίσης θα πρέπει να ε, ευθυγραμμίσουν την εξωτερική τους πολιτική με την εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Ε, σήμερα είναι 10η Ιανουαρίου όπου η Σερβία ε, γιορτάζει μια εορτή που έχει απαγορευτεί από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Βοσνίας Ερζεχοβίνης και ο πρόεδρος επισκέφτεται την Σερβία που σημαίνει ότι κάθε ευρωπαϊκού τύπου δραστηριότητα αντισταθμίζεται από μια ρωσική, μάλλον φιλορωσική δραστηριότητα. Η Σερβία δεν θα πρέπει να διακινδυνεύσει τη θέση της σε σχέση με την Ένωση και είναι απαραίτητο να καταγγείλει σαφώς τις απόψεις του κύριου Ντόντικ και πιστεύω και ελπίζω πως αυτό θα γίνει και ότι θα υπάρξει, πρόοδο πρόοδος πραγματικά. Κάποια ανοιχτά ζητήματα σε σχέση με την Κροατία είπαμε ήδη ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις διμερείς ε, σχέσεις και να τις έχουμε στο μυαλό μας. Θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό, γιατί αν δεν λυθούν τα προβλήματα του παρελθόντος, η Σερβία δεν θα μπορέσει να προοδεύσει. Θα πρέπει λοιπόν να επιληθούν τα ανοιχτά διμερεί ζητήματα. For his excellent works, ε, as always. I think all areas in... Ο κύριος Δέλη. Ευχαριστώ. Εξαιρετική εργασία του εισηγητή. Καλύπτονται όλα τα ζητήματα. Είναι πολύ ισορροπημένο το κείμενο και αποτελεί πολύ καλό πλαίσιο για τη μελλοντική μας εργασία εδώ. Θέλω να δεν επενέσω το γεγονός ότι Υπάρχει μια αναφορά στις εθνικές μειονότητες ήδη στο σχέδιο και αυτή είναι πολύ καλή αρχή και πολύ καλό σημάδι για όλους τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Πέρα από το θέμα των μειονοτήτων, να καλωσορίσω επίσης τη δέσμευση της Σερβικής Κυβέρνησης για οικονομικές μεταρρυθμίσεις που έχουν αρχίσει να δείχνουν αποτελέσματα, αλλά πέρα από την γενική μακροοικονομική εικόνα θα ήθελα να δοθεί περισσότερη προσοχή στις μικρομεσαίες και στους επιχειρηματίες και άρα οι τροπολογίες μας θα εστιάσουν σε αυτό το στοιχείο κυρίως και προσβλέπω σε συνεργασία με το γραφείο του κ. Μακάλιστερ για αυτό το θέμα και μια γενικότερη παρατήρηση. Ο πρόεδρος Μπρόκ είπε νωρίτερα ότι ε, ο δρόμος της Σερβίας προς την Ένωση είναι πολύ σημαντική και ο καλός ρυθμός διαπραγματεύσεις είναι σημαντικός και η Σλοβακική Προεδρία πέρυσι έδωσε όση όθεση μπορούσε ώστε να διατηρηθεί αυτός ο καλός ρυθμός. Ελπίζω πραγματικά ότι η Μάλτα και η Αστονία θα διατηρήσουν ε, αυτό το ρυθμό στις διαπραγματεύσεις και ότι το κοινοβούλιο μας θα πρέπει να επιμείνει για να διατηρηθεί ψηλά στην ημερήσια διάταξη της Προεδρίας ε, η Σερβία και φέτος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πέτερ. E, Ευχαριστώ. Ο κύριος να ε, γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση στη Σερβία και έχει αφιερώσει πολλή προσπάθεια ώστε η Σερβία να προχωρήσει στο δρόμο προς την Ένωση και γι' αυτό θέλω να το ρωτήσω, να το ζητήσω μάλλον να βοηθήσει στην επίλυση του θέματος του σερβικού νόμου για τις ε, αρμοδιότητες του των κρατικών οργανισμών όσον αφορά τα εγκλήματα πολέμου. Έχω τονίσει το θέμα αυτό επανειλημμένως. Η Σερβία έχει πάρει το δρόμο για το δικαστήριο της Χάγης. Μεγάλη απειλή για τους βετεράνους της Κροατίας, αλλά είναι απειλή και για άλλες χώρες που δεν είναι μέλη της Ένωσης, όπως το Κωσυφοπαίδιο, διότι βασίζεται σε αυτό το νόμο που αναφέρει, επί με βάση το οποίο συνελήφθη ο κ. στη Γαλλία και ε, τα, τα, το οποίο κάποια άρθρα πρέπει να διαγραφούν. Ε, ε, Εγώ ανησυχώ πολύ όσον αφορά την έλλειψη προόδου στον τομέα του σεβασμού των, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στη παιδεία και αναφέρομαι εδώ στην κροατική εθνική μειονότητα στη Σερβία. Α, λυπούμε που ο Γενικός Εισαγγελέας ε, του, του Δικαστηρίου της Χάγης καθώς και ο πρόεδρος της Χάγης είπαν ότι η Σερβία δεν συνεργάζεται με το δικαστήριο και αυτό οδηγεί στην ριζοσπαστικοποίηση του πολιτικού προσκυνείου της χώρας. Να τονίσω και να προσθέσω ότι η Ρωσία έχει πολύ έντονη ε, επιρροή, είναι ιδιαίτερα παρούσα και πιστεύω πως η Σερβία θα πρέπει να απομακρυνθεί από την Ρωσία διαφορετικά δεν θα μπορέσει να μπει στην Ένωση. Και επίση ε, καταδικάζω τις στρατιωτικέ ασκήσει στα σύνορα. Ευχαριστώ, Μπόγκοβιτ. Ευχαριστώ, κύριε και εγώ είμαι μέρο τη αντιπροσωπεία με τη Σερβία, γι' αυτό λαμβάνω τον λόγο. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή. Πέρσι πήγα διάφορε φορέ στη Σερβία, γνωρίζω πολύ καλά τα θέματα αυτά. Ξέρω ότι ο εισηγητής έχει βάλει πολύ προσπάθεια σε αυτή την έκθεση, έχει επισημάνει σωστά ότι πρέπει να επισημανθεί και έχει επικρίνει αυτά που πρέπει να επικριθούν. Έχουμε καλύψει λοιπόν όλα τα βασικά στοιχεία. Να υπογραμμίσω επίση αυτή την έκθεση ότι εγώ παρακολουθώ την οικονομική κατάσταση στη Σερβία, έχει βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Πρέπει όμως να είμαστε και πιο ρεαλιστές αν λάβουμε υπόψη και τη δημογραφική εξέλιξη στη Σερβία. γεννήσεις είναι πολύ λιγότερες οι γεννήσεις από τους θανάτους στην Σερβία και αυτό δείχνει τη σημασία του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Σερβία. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει τη Σερβία να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα ώστε να προληφθούν αυτά τα προβλήματα και να μπορέσει να υπάρξει μια ειρηνική εξέλιξη στη Σερβία. Επίσης να υπογραμμίσουμε και το ρόλο που μπορεί να παίξει η Σερβία ως σταθεροποιητικός παράγων στη γειτονιά της. Αναφέρθηκε επίσης και η προσέγγιση με τη Ρωσία και η επιρροή της. Πρέπει να έχουμε σαφείς ιδέες για το πώς θα ενισχύσουμε το ρόλο της Σερβίας και η διαδικασία της ε, ένταξης θα πρέπει να είναι ελκυστική για τους πολίτες της Σερβίας. Κάποια κράτη-μέλη θέλουν να βγουν τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο ο ενθουσιασμό στη Σερβία για την ένταξή τη έχει μειωθεί και κιόλα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Θα δώσω το λόγο στην κυρία. Πώ την είπε, Καλαβέρα. Δεν άκουσα. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για το σχέδιο αυτό έκθεση, το σχέδιο αυτό ψηφίσματο. Συμφωνούμε με τη γενικότερη αξιολόγηση και καλωσορίζουμε το σχέδιο της έκτασης που θεωρούμε ότι είναι ισορροπημένη. ορίζουμε όπως και εσεί την ε, πρόοδο της Σερβίας. Και χρειάζονται στρατηγικοί στόχοι σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση πρέπει να σας πούμε ότι γενικά είμαστε ικανοποιημένοι σε ό,τι αφορά τα σκέλη αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ε, εκτιμά ιδιαίτερα τι προσπάθειε της Σερβίας για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Και δίνουμε χρηματοδοτική βοήθεια σε ό,τι αφορά τη Σερβία για τις ε, ανάγκες που έχει, σε ό,τι αφορά την ε, προσχώρηση είμαστε σε καλό δρόμο με τι διαπραγματεύσει. Έξι κεφάλαια ανοιχτά. Ένα προσωρινά έχει ήδη κλείσει. Και τι χρειαζόμαστε πλέον. Μία νέα δέσμευση από πλευρά τη Σερβία για να προχωρήσει με τι μεταρρυθμίσει. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την, το δικαστικό, την καταπολέμηση της διαφθοράς, ελευθερίας, έκφρασης, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, μεταρρύθμιση της ε, δημοσίας και ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Εξίσου σημαντικά είναι τα θέματα της πρόοδου για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου. Και επίσης η Σερβία θα πρέπει να συνεχίσει με την ε, εναρμόνιση με το κοινωτικό κεκτημένο σε ό,τι αφορά το άσυλο και άλλα θέματα. Ελπίζουμε ότι η σταθερή πρόοδο στους τομείς αυτούς θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν να ανοίξουν και άλλα κεφάλαια διαπραγματεύσεις το 2017. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προελιάνει το έδαφος και είμαστε δεσμευμένοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη Σερβία και οικονομικά αλλά και από πλευρά τεχνογνωσίας σε αυτή τη διαδικασία προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχει ο κ. Μακάλιστερ, ο εισηγητής. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσω ιδιαίτερος για τις ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις όχι μόνο των ε, σκιωδών αλλά και των άλλων συναδέλφων και χαίρομαι ιδιαίτερα που ήταν τόσο επικοδομητική συζήτηση Μέχρι 18 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι έχουμε χρόνο για την υποβολή τροπολογίων και θεωρώ δεδομένου ότι θα καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη λογική δεύτερη ανάγνωση και όπως προγραμματίζεται θα ολοκληρώσουμε όλα στο Στρασβούργο. Φαίνεται ότι όλοι συμφωνούμε ότι είναι σε καλό δρόμο η Σερβία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασφαλώς πολλά ακόμα θα πρέπει να γίνουν, αλλά νομίζω ότι όλοι από όλο το πολιτικό φάσμα ε, έχουμε συμφέρον να υποστηρίξουμε τη Σερβία και θεωρώ ότι πρόκειται για ένα ε, τεράστια σημασία πολιτισμικό κράτος ε, με πολιτισμική κληρονομιά και θεωρώ ότι θα αποτελούσε αυτό, μάλλον η ένταξη θα αποτελούσε εμπλουτισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 18 Ιανουαρίου στις 12 η ώρα. Μπορούμε να κλείσουμε λοιπόν αυτό το σημείο και περνάμε στην πρώτη εξέταση της έκθεσης 2017 για το Κοσμοπέδιο με την κυρία Λούνα Τσέκος, εισηγήτρια. Σας υπενθυμίζω ότι όπως και για τη Σερβία είχαμε δει την παρουσίαση του, τον Νοέμβριο από τον Επίτροπο Χαν του πακέτου για την ε, ένταξη, για την ε, πρόθεση της ένταξης. Το Μάιο πρότεινε Κομισιόν φιλελευθεροποίηση προξενικών ε, θεωρήσεων για το κοσυφοπαίδιο. Ακόμα εκκρεμούν ορισμένε βασικέ προποθέσει, αλλά θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Λούνα Τσέκ για να παρουσιάσει τη θέση τη για τι τροπολογίε και την εκθεσή τη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω όμως αγγλικά παρόλα αυτά. Και εγώ θέλω να ξεκινήσω με τα θετικά πράγματα που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό για το κόσμο Πέδιο που είναι τμήματα της έκθεσής μου. Καταρχήν η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με το κόσμο Πέδιο που ετέθη σε εφαρμογή την 1η Απριλίου, η πρώτη συμβατική σχέση που δημιουργείται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη πιο νέας ευρωπαϊκής χώρας. Στις 11 Νοεμβρίου ήμουν μαζί με τον Επίτροπο Χάν στην Πριστίνα και ήμασταν παρόντες στην εκκίνηση της Ευρωπαϊκής Ατζέντα Μεταρρύθμισης που είναι η προσπάθεια να εφαρμοστούν όλα αυτά που βρίσκονται στη Συμφωνία Σύνδεσης και Σταθεροποίησης και εκεί και το Κοσφοπέδε πρέπει να δείξει σαφή πολιτική θέληση και αποφασιστικότητα για την εφαρμογή όλων των πτυχών του οδικού χάρτη. Αυτή η συμφωνία σύνδεση και σταθεροποίηση θα υποστηρίξει του πολίτε του Κωσυφοπαιδίου, πεδίου, ιδίω σε ό,τι αφορά τη βελτίωση τη οικονομική του κατάσταση, τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και όλα αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι έχουν περισσότερη σχέση με το κράτο του και με την διατήρηση με την, παρου... την συνέχιση της παρουσίας του στο Κωσυφοπέδιο. Δεύτερο στοιχείο ήταν η υπογραφή της Συμφωνίας Πλαισίου για τη συμμετοχή του κωσφοπεδίου στα ευρωπαϊκά προγράμματα <clears throat> και τέλο υπήρξε η Συμφωνία για το Διάλογο για ένα ανεξάρτητο τηλεφωνικό κωδικό για το κοσφοπέδιο δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως ακόμα, αλλά σύντομα οι πολίτες του κοσφοπεδίου θα μπορούν να έχουν ένα αυτόνομο κωδικό και όχι να γίνεται η πρόσβαση με Σλοβενίας ή άλλων χωρών. Τέλος, έχουμε ακόμα το <coughs> εκρεμές πράσινο φως της Κομισιόν για τη φιλελευθεροποίηση των προξενικών θεωρήσεων που εξαρτάται από δύο ακόμα προαπαιτούμενα. Είναι το Κοσμοπέδιο η μόνη χώρα από τις έξι υποψήφιες χώρες της, ε, ε, των Δυτικών Βαλκανίων που οι πολίτε τη δεν μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα για τι μήνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και χαίρομαι λοιπόν όταν δόθηκε το πράσινο φω από την Κομισιόν. Αυτή τη στιγμή το μπαλάκι είναι στο γήπεδο του Κωσυφοπεδίου. Υπάρχουν δύο προαπαιτούμενα το θέμα των συνόρων, της οριοθέτησης των συνόρων με το Μαυροβούνιο πρέπει να εγκριθούν από το Κοινοβούλιο του Κωσυφοπεδίου. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες και <clears throat> διαμάχες για το θέμα αυτό, αλλά ξέρουμε ότι πρέπει τώρα το Κωσυφοπεδίο να το κάνει, γιατί έχει υπογράψει αυτή η συμφωνία το, η κυβέρνηση του Κωσυφοπεδίου. Αν θέλει το Κωσυφοπεδίο να χρησιμοποιήσει αυτό το πράσινο φως από την Κομισιόν, τότε πρέπει πράγματι να εκπληρώσει τα προαπαιτούμενα και επίσης το ίδιο αφορά για αυτούς για τους ε, υψηλά ειστάμενους που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα και διαφθορά και εκεί πρέπει να δράσει η κυβέρνηση και τότε θα μπορέσουν να εξασφαλιστούν τα προαπαιτούμενα για την ελεύθερη διακίνηση και την άρση των, της υποχρέωσης προξενικής θεώρησης. Αλλά είναι σαφές ότι το κολυφοπέδιο πρέπει να επιτύχει αυτά τα προαπαιτούμενα. Λυπάμαι επίση και το λέω στην έκθεσή μου για την πόλωση που έχει δημιουργηθεί και ελπίζω θα μπορέσουν να βελτιωθούν τα πράγματα το 2017. Υπάρχουν και άλλα θετικά πράγματα όπως η συμφωνία για την για τον διάλογο στα δικαστικά θέματα μεταξύ Κωσυφοπεδίου και Σέρβία, αλλά αυτό πρέπει να εφαρμοστεί και σε άλλε πτυχέ του διαλόγου. Το είπαμε και στην έκθεση για τη Σερβία. Ο διάλογο αυτό μεταξύ των δύο μερών είναι μια πάρα πολύ θετική διαδικασία. Θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Μογερίνη και το προσωπικό του για το, την υποστήριξή του και την υποστήριξη των πρεσβειών και τη Ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία εκεί, αλλά η εφαρμογή πρέπει να γίνει από τι αρμόδιε αρχέ και την κυβέρνηση, αλλιώ δεν θα επιτευχθεί τίποτα. Ένα άλλο σημείο που ανέφεραν τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα δικαιώματα των γυναικών, το θέμα αντιμετώπιση τη οικιακή βία που εξακολουθεί να είναι μεγάλο θέμα στο Κωσυφοπαίδιο, όχι φυσικά μόνο στο κοσφοπέδιο και σε άλλε χώρε τη περιοχή, αλλά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόβλημα, αλλά θέλω να το τονίσω και στην εκθεσή μου. Η κατάσταση των ΛΟΑΔ έχει βελτιωθεί, υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, αλλά ακόμα εξακολουθεί να υπάρχει φόβος και μια αίσθηση καταπίεσης. Το, κατά, το κράτος δικαίου, αγώνας κατά της διαφθοράς πρέπει να αντιμετωπιστούν και πρέπει να υπάρξει για ένα άλλο θέμα και μια τροποποίηση της ενεργειακής στρατηγικής. Χρειάζεται το κοσμοπέδιο να έχει μια ενεργειακή στρατηγική που να οδηγήσει στην εν καιρό εγκατάλειψη των ε, ορυκτών καυσίμων ε, ο λιγνής που χρησιμοποιείται δημιουργεί προβλήματα υγείας. Πρέπει να αυξήσουμε λοιπόν και την διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και την αποτελεσματικότητα στην χρήση της ενέργειας. Και στην έκθεσή μου, φυσικά, όπω το κάνω εδώ και πολλά χρόνια, ζητώ από τα πέντε κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν αναγνωρίσει το κοσμοπέδιο να προχωρήσουν στην αναγνώριση. Πολλέ από αυτέ τι πέντε χώρε εργάζονται στενά με το κοσμοπέδιο σε πολλά επίπεδα δίνουν ακόμα και βίζες για τις χώρες του Σέγγεν. Αναγνωρίζουν λοιπόν τα διαβατήρια του Κωσυφοπεδίου, αλλά δεν το αναγνωρίζουν ω χώρα σε διεθνέ επίπεδο. ήταν πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν για να μπορέσει το Κωσυφοπέδιο να συμμετέχει και σε μεγαλύτερα και περισσότερα διεθνή φόρα. Σα υπενθυμίζω, το Κωσυφοπέδιο έχει ήδη αναγνωριστεί από 113 από τι 193 χώρε του ΟΗΕ. Εν κατακλείδη, να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία και το δικό μου προσωπικό και την ομάδα μου για την υποστήριξη που μου έδωσαν και προσβλέπω σε συνεργασία με τους χειοδησίγητες που έχουμε ήδη συνεργαστεί υποφελώς και στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Περνάμε με τους σκιώδεις εισηγητές, ο κύριος Αλάτουσον. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Λουνατσέκ. Να ευχαριστήσω την κυρία Λούνατσεκ λοιπόν για την πάρα πολύ επαγγελματική δουλειά που έκανε και πολύ ισορροπημένη η έκθεση της. Περιλαμβάνει λοιπόν η έκθεση όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κοσίφου πεδίου. Αντί λοιπόν να επικεντρωθώ σε αυτά που ήδη περιλαμβάνονται στην έκθεση, επιτρέψτε μου να εκφράσω κάποια ζητήματα που απασχολούν την ομάδα του ΕΛΚ. Το σχέδιο έκθεση αναφέρεται εν συντομία στην οικονομική κατάσταση που του κρατεί στη χώρα. Και παρά το γεγονός ότι συμφωνώ με την χαρά που εκφράζει η συγγήτρια για τα μεγαλύτερα φορολογικά έσοδα, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η βάση της ε, οικονομίας μιας χώρας δεν είναι η δυνατότητα συλλογή φορών, αλλά η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα στην παράγραφο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ξέρω ότι η συγκεντρία μίλησε για βία ή τρομοκρατία. Καθίστε σαφέ στην παράγραφο ότι το πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση είναι ο ακραίος Ισλαμισμός. Και θα υποβάλει ε, τροπολογία το ΕΛΚ για να κατανοήσουμε καλύτερα το πρόβλημα, γιατί πιστεύουμε ότι έτσι θα πετύχουμε καλύτερες λύσεις μία συγκεκριμένη πρόταση θα ήταν το πώς ε, θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τη χρηματοδότηση προς ε, τρομοκρατικές ε, οργανώσεις από χώρες όπως η Ειδική Αραβία και το Κατάρ. Τέλος, να σχολιάσω τις όχι και τόσο φυσιολογικές σχέσεις μεταξύ Σερβίας και Κωσικοπεδίου. Η σύλληψη του πρώην Πρωθυπουργού Χαρδινάη, θεωρούμε ότι βάζει ερωτηματικά σε ό,τι αφορά και τις αποφάσεις του δικαστηρίου για τα εγκλήματα στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Ό,τι συνέπειες και αν έχει αυτό προσωπικά για τον κύριο Χαρδινάη. Νομίζω ότι η Σερβία είναι αυτή που έχει να χάσει τα πιο πολλά από το περιστατικό αυτό. Γιατί πολλοί διαπιστώνω ότι όλα αυτά τα συμβαίνουν στο κενό. Ο πόρεμος Μητροβίτσα, η αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά το δικαστικό σώμα, οι απειλές για τη μονομερή ίδρυση σε ό,τι αφορά α, κάποιες ε, κοινότητες στη Σερβία αποτελούν ε, παραδείγματα και επίσης ε, και η άρνηση το να γίνει θρησκευτικό εορτασμό των Χριστουγέννων, ούτε είναι, αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό σημείο. Είμαστε αισιόδοξοι για τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις και ελπίζουμε να είναι τουλάχιστον όσο επικοδομητικές όσο και πέρσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Μπενιφέη, ο οποίος θα μιλήσει εξ του κύριου Παντσέρη. Στο όνομα του σκιώδου εισηγητή μας, του Αντώνιο Μπαντζέρη, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Λούνατζεκ για την εξαιρετική της εργασία. Το σχέδιο έκθεσης που μας υπέβαλε λαμβάνει υπόψη τις βασικές ανησυχίες ε, πολιτικού τύπου όσον αφορά το Κωσυφοπέδιο. Η έναρξη ισχύω τη Συμφωνία Σταθεροποίηση και Σύνδεση Ένωση Κοσμοπεδίου 1η Τετάρτου 2016 είναι ένα αποφασιστικό βήμα για την ένταξη ε, του κοσμοπεδίου στην Ένωση και το σχέδιο μεταρρύθμισης αποτελεί ε, μια θετική εξέλιξη, θα είναι μια βάση για να ε, παγιωθεί η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ε, η πόλωση, η μόνιμη πόλωση του πολιτικού προσκυνείου, η ανάγκη συνεργασίας για την επίτευξη συμφωνιών διώσιμων ε, στην πορεία προς την Ευρώπη και απελευθέρωση των θεωρήσεων ως βασικό βήμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Γι' αυτό όμως ανησυχούμε όσον αφορά την τελμάτωση στην κοινοβούλη, όσον αφορά την επικύρωση της συμφωνίας ορίων με το Μαυροβούνιο. Η απελευθέρωση των θεωρήσεων θα μπορέσει να δοθεί μόνο αν το κοσφοπέδιο έχει τηρήσει όλα τα κριτήρια, μεταξύ αυτών και οι συμφωνίες ε, υψηλού επίπεδου για την διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. Για το σερβικά σύνορα είναι σε απαραίτητο το κοσφοπέδιο να συμφωνήσει στη συμφω... Ε, στο πλαίσιο τη συμφωνίας που έχουμε φτιάξει με την Ένωση και ε, με βάση την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Χωρί να μπούμε σε όλε τι λεπτομέρειε, οι σοσιαλιστέ θα στηρίξουν τη γενική προσέγγιση. Ο δυσκιώδη μα εισηγητή ε, Παντζέρη θα υποβάλει κάποιε τροπολογίε, ε, προσέχοντα πρώτα την καταπολέμηση του διαφθορά και του οργανωμένου εγκλήματο και την ανάγκη συντονισμού ανάμεσα στου θεσμού που εντοπίζουν, ερευνούν και διώκουν τι υποθέσει διαφθορά. Δεύτερον, την ανάγκη για αποτελεσματικά προγράμματα ώστε να αντιμετωπιστεί η οι βίες ακρότητες και η ριζοσπαστικοποίηση και, ε, θα προαχθεί έτσι ο διάλογος. Είναι σημαντικό να δοθεί μεγαλύτερη πολιτική σημασία και συνεργασία ανάμεσα στα τμήματα της κυβέρνησης για να επιτευχθούν ε, ε, πρόοδοι, να αξιολογηθούν οι προκλήσεις επί τη βάση της αξιολόγησης ε, που θα έχουμε ε, για τα σχολεία και τις σχέσεις ανάμεσα στους ε, εκπαιδευτές και τους μαθητές. επίτε, επίσης, επιθεωρήσεις εργασίας και ε, ειρηνοδικία, ώστε οι πολιτικές και οι νομοθεσίες θα έχουν ενημερωθεί και ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται από το, τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας να ξεπεραστούν. Ευχαριστήσω ακόμα μια φορά στο όνομα του κυρίου Παντζέρη την κυρία Τσεκ και την επόμενη εβδομάδα θα δουλέψουμε για πιθανέ συμβαστικέ. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριο Μακάλιστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λούνατσεκ για την ε, πλήρη και περιστατωμένη έκθεσή της για το Κωσυφοπαίδιο. Θέλω να χαιρετήσω όχι μόνο το Κοσμοπεδίο αλλά και τη Σερβία στην προσήλωση για να υπάρξει ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ τους και τις προσπάθειές τους για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις συμφωνίες που έγιναν με τη διαμεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι πια είναι καιρός να προχωρήσουμε στην πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών που έχουν ήδη επιτευχθεί με καλή πίστη και ιδίως εγκαίρως. Και θέλω επίση να ενθαρρύνω και τι δύο πλευρέ, και το Κωσυφοπέδιο και τη Σερβία, να βρουν νέου χώρου διαλόγου, νέα θέματα διαλόγου, για να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών τους και να υπάρξει μια πλήρης ομαλοποίηση των σχέσεών τους. Ζητώ από την Υπηρεσία Εξωτερικής δάση να κάνει μια αξιολόγηση της επίδοσης και των δύο πλευρών στην επίτευξη αυτών των υποχρεώσεων. Ο κ. Πίκουλα. Ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ και εγώ την κυρία Λούνατσεκ για την πολύ καλή έκθεσή τη, η οποία παρουσιάζει με αντικειμενικό τρόπο την κατάσταση στο κοσμοπέδιο και αυτά τα οποία έχουν επιτευχθεί και τι ευκαιρίε οι οποίε έχουν χαθεί. Το πιο σημαντικό βέβαια ήταν η Συμφωνία σύνδεση και σταθεροποίηση και η έναρξη του θεματολογίου μεταρρυθμίσεων καθώ και οι συστάσει για την ε, φιλελευθεροποίηση των προξενικών θεωρήσεων. Αυτό ναι, δεν έχει επιτευχθεί ακόμα γιατί υπάρχουν δύο προαπαιτούμενα που δεν επιτεύθησαν. Όπως ελέγχθη, η οριοθέτηση του συνόρου με το Μαυροβούνιο. Ξέρουμε όμως ποιες είναι οι επιτόπιες συνθήκες. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να επιτευχθούν τα δύο προαπαιτούμενα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να ακυρώσει αυτή την απόφαση και να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία για τους πολίτες του Κοσφοπεδίου. Ως ε, πρόεδρος της αντιπροσωπείας ε, και για τη συνεργασία με το Κοσφοπέδιο πρέπει να πω ότι και η αντιπροσωπεία μας λειτουργήσε πολύ καλά. Όλα τα μέλη έχουν συμβάλει στις δύο συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν εγκρίναμε το νοδικό χάρτη και τις συστάσεις και πρέπει να υπογραμμίσω επίσης και τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ στις σχέσεις Κωσυφοπεδίου και Σερβίας. Έχουμε τον ενιαίο κωδικό για το Κωσυφοπέδιο, έχουμε το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά εξακολουθεί το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά υψηλού να είναι προβλήματα όπως και η έλλειψη ελευθερίας στα μέσα ενημέρωσης. Όλα αυτά είναι προσκόμματα για την ένταξη του κοσυφοπεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω ότι η Συμφωνία Σταθεροποίησης και σύνδεση θα είναι το πρώτο βήμα που θα οδηγήσει και σε περαιτέρω νέα θετικά μηνύματα για τη νεότερη αυτή χώρα της, Ευρωπαϊκής, της Ευρώπης που θα υποστηρίξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι και. Ευχαριστώ. Η κυρία Λεούνατσεκ μίλησε για θέματα που υπάρχουν στο κοσυφοπέδιο, αλλά θεωρώ ότι η πραγματική κατάσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη στο κοσυφοπέδιο από ότι αυτοί που απεικονίζεται στην έκθεση. Ας ξεκινήσουμε με τα τυπικά θέματα. Υπάρχει μια παραλληλισμός μεταξύ κοσυφοπέδιου και Κρυμαία. Και θεωρούμε ότι η ανεξαρτησία στο κωσυφοπέδιο προλύανε την ανεξαρτησία στην Κρυμαία. Αλλά το θέμα είναι, η διαφορά είναι ότι η Κρυμαία θα μπορούσε να είναι ανεξάρτητο κράτο. Αλλά το κωσυφοπέδιο είναι τεχνητό κράτο, το οποίο το υποστηρίζει η διεθνή κοινότητα και οι Αμερικάνοι. Φυσικά η Κρυμαία έχει δικαίωμα να μπει στη Ρωσική Ομοσπονδία, όπω και το 25 μπορεί να μπει στην Ευρωπαϊκή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η πραγματική κατάσταση στο κοσμοπέδιο είναι πάρα πολύ επικίνδυνη σε ό,τι αφορά δηλαδή την προσχώρηση της, του κοσυφοπαίδιου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πιστεύω ότι είναι εντεχνία του κ. Πέτερλε. Η κυρία Λούνατσακ είναι πάρα πολύ αξιόπιστη ως εισηγήτρια και θα ήθελα πραγματικά να τη συγχαρώ για την ε, και χαίρομαι που και στην περίπτωση του κοσφοπεδίου μιλάμε για πρόοδο. Και εδώ τα στατιστικά στοιχεία είναι α, θετικά. Δέκα φορές, σε δέκα περιπτώσεις ε, καλωσορίζουμε την πρόοδο, σε τέσσερις περιπτώσεις εκφράζουμε ανησυχία και σε δέκα περιπτώσεις κάνουμε προτάσεις. Το θέμα, ξέρετε, είναι και θέμα πολιτικής κουλτούρας, ότι αφορά το να υπάρχει μια διάθεση να γίνουν δεκτές οι ιδέες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ισχύει και για τη Σερβία προφανώς. Και ίσως να είναι δύσκολο να υιοθετηθούν τα ευρωπαϊκά στάνταρα, αλλά ελπίζω να το πετύχει αυτό η Σερβία για το κοσμοπέδιο. Ευχαριστώ κυρία Φαγιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρα και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους, ε, τη συνάδελφο την εισηγήτρια κυρία Λούνατσεκ. Πάντα με μεγάλη χαρά συνεργάζομαι μαζί τη και πραγματικά ε, είναι προσδεκτή η δέσμευσή τη να βοηθήσει το κοσυφοπαίδιο. Αναφέρθηκαν ε, διάφορα θετικά στοιχεία για το 25, δεν θα τα επαναλάβω. Θα ήθελα να περιοριστώ σε ένα θέμα, το καθεστώς απελευθέρωση από τις θεωρήσεις για το κοσυφοπαίδιο και συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι αυτό αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα για τους πολίτες. Και λυπάμαι που δεν σημειώθηκε πρόοδο στο θέμα αυτό του τελευταίου μήνε. Σίγουρα το μπαλάκι πλέον είναι από, από την πλευρά της του κοσυφοπεδίου. Να σας πω ότι καταβάλαμε πάρα πολλέ προσπάθειες για να βοηθήσουμε τις αρχές του κοσυφοπεδίου προκειμένου να πληρώσουν τις τελευταίες δύο όρους για το Μαυροβούνιο, για την επικρίση της σχετικής συμφωνίας και το θέμα της καταπολέμησης της διαφθοράς. Κατανοώ τις ευαισθησίες που εμπεριέχονται σε θέματα διαχείρισης των συνόρων, αλλά θα ήθελα να καλέσω εκ νέου τις αρχές του Κωσυφοπέδιου να επιταχύνει τη διαδικασία αυτή, γιατί έχουμε μια ευκαιρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προχωρήσουμε και ελπίζω να την αξιοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή, γιατί όπω σα είπα, αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο ιδιαίτερα σε του νέου. Να ανοίξει δηλαδή η πόρτα για ένα καθεστώ ελεύθερο από τι θεωρήσει και μια μεγαλύτερη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε Κούκαν. Ευχαριστώ. Και εγώ να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερω την έκθεση τη κυρία Λούνα, της έκθεσης Πάρα πολύ καλή έκθεση, πραγματικά. Και την εκτιμώ ιδιαίτερω είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ελπίζω το 2017 να συνεχίσει το Κοσφοπέδιο να κινείται προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντίθεση με κάποιους προηγούμενους ομιλητές. Ακούσαμε διάφορα στοιχεία και θα ήθελα να τονίσω ότι ήταν μεγάλη επιτυχία η θέση σε ε, εφαρμογή, σε ισχύ του SAA τη συμφωνία σταθεροποίηση. Τα σύνορα με το Μαυροβούνιο. Θα πρέπει να επιληθεί το θέμα αυτό, η γραμμή δηλαδή, με το Μαυροβούνιο, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με την απελευθέρωση του κατέσταση των θεωρήσεων. Κατά πολέμηση επίσης της διαφθοράς, προκειμένου να υπάρχει αξιοπιστία. Αυτό προϋποθέτει πολιτική βούληση και ελπίζω να επιδείξουν η ηγεσία οι αξιωματούχοι της, του οικοσκοπεδίου και θα ήθελα όπως και στην περίπτωση της Σερβίας να καλέσω και τους αξιωματούχους του οικοσκοπεδίου να συνεχίσουν το διάλογο μεταξύ Βελεγραδίου και Πρίστινα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνω το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λούνατσεκ, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, ιδιαίτερα την εισηγήτρια, για το σχέδιο εκθεσή σας για το κοσφοπέδιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται τις ε, εκτιμήσεις σας για το Κωσυφοπαίδιο και εμείς ανησυχούμε για την πολιτική κατάσταση στην ε, Πριστίνα. Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχουν σημαντικές αποφάσεις οι οποίες εκκρεμούν οριοθέτηση των συνόρων με το, ε, με το Μαυροβούνιο και η σχέση με τις ε, σε, πλειοψηφίας ε, κοινότητες και δήμους. Πρέπει επίσης να εστιάσει περισσότερο στις μεταρρυθμίσεις στο Κοσμοπέδιο ώστε να μπορέσει να έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον τρόπο αυτό θα εκμεταλλευτεί και τις ευκαιρίες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με την θέση εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Τώρα έχουμε ένα πλήρες πλαίσιο για πιο στενό πολιτικό διάλογο και εμβάθυνση των οικονομικών μας σχέσεων και θα πρέπει να αντλήσουμε το μέγιστο όφελος από αυτά. Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει από την κυβέρνηση του Κωσυφοπεδίου και την Κομισιόν είναι εργαλείο για να μπορέσει το Κωσυφοπέδιο να μεγιστοποίηση τα ωφέλη αυτής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης και ελπίζουμε ότι το Κοσμοπέδιο με σαφής ενέργειας θα καταδείξει ότι υποστηρίζει αυτό το θεματολόγιο και θα κάνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Για τη φιλελευθεροποίηση θεωρήσεων πρέπει το Κοσμοπέδιο να κυρώσει τη συμφωνία των συνόρων με το Μαυροβούριο και να συνεχίσει τον αγώνα κατά της διαφοράς και του οργανωμένου εγκλήματος ώστε να γίνει πραγματικότητα η φιλελευθερωποίηση για τις βίζες και για το λαό του Κωσυφοπέδιου. Επίσης έχουμε την συμφωνία πλαίσιο που θα επιτρέψει το Κωσυφοπέδιο να συμμετάσχει σε μια σειρά από ευρωπαϊκά προγράμματα και έτσι θα διευρύνει τις ε, σχέσεις και τη σύνδεση μεταξύ των κοινωνιών του Κωσυφοπεδίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η χρηματοδότηση θα φτάσει να, το ευρύτερο να το φάσμα στρωμάτων της κοινωνίας στο Κωσυφοπέδιο. Γι' αυτό θα παραμείνουμε προσιλωμένοι στην προσπάθεια αυτή να προωθήσουμε το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο του Κωσυφοπεδίου το 2017. Ευχαριστώ πολύ με την άδεια της εισηγήτριας θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Σουίτσα, την οποία η... που δεν μπορούσα να της δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή είμαι και αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Κωσυφοπαίδιο, θα ήθελα να πω ότι και εγώ ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για το θέμα αυτό. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να πω. Οι περισσότεροι από εμά συμφωνήσαν σε σχέση με την κατάσταση του Κωσυφοπαίδιου Θέλω να συγχαρώ την κυρία Λούνατσερ για την εξαίρετη και τόσο επαγγελματική έκθεσή της και για την δέσμευσή της για την πρόοδο στο κοσμοπέδιο. Έγιναν κάποιες θετικές ενέργειες όπως η υπογραφή της συμφωνίας ε, σύνδεσης και σταθεροποίησης και το θεματολόγιο μεταρρύθμισης, ε, η δημιουργία ενιαίου τηλεφωνικού κωδικού για το κοσυφοπαίδιο. Βέβαια δεν προχώρησε η φιλελευθερωποίηση για τι προξενικές θεωρήσεις σε λήψη δύο προαπαιτουμένων. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο τώρα να ακυρωθεί μια συμφωνία για το νοριοθέτηση των συνόρων με το Μαυροβούνιο, αλλά αυτό θα πρέπει να παραμείνει ένα από τα προαπαιτούμενα και χαίρομαι που ζητάτε από τα πέντε κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν αναγνωρίσει το κοσμοπέδιο να το κάνουν. Το Ευρωπαϊκό, το Συμβούλιο Μάνα τη Ευρώπη έχει προσκαλέσει το Κωσυφοπαίδιο να γίνει παρατηρητή στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και αυτό είναι μια άλλη μορφή αναγνώρισης για το Κωσυφοπαίδιο και μια πρόσκληση να συμμετάσχει στα ευρωπαϊκά τεχθενόμενα και υπογραμμίζω την ανάγκη να υπάρξει πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας που έχει κάνει το Κωσυφοπαίδιο με τη Σερβία και αυτό είναι απαραίτητο να να μειωθεί η πόλωση στο εσωτερικό του κοσφοπεδίου για να προωθεί το μέλλον του. Ευχαριστώ η κυρία Λούνατσεκ και εγώ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές ε, και όσους ήταν στην αποστολή, αλλά και τους συναδέλφους που στηρίζουν την πορεία του Κωσυφοπεδίου προς την Ένωση και που στηρίζουν όλους όσους θέλουν αυτή η χώρα να προχωρήσει και να αποτελέσει κομμάτι περισσότερο αυτής της κοινή Ευρώπης. Ε, εγώ προσλάβω σε όλες αυτές τις τροπολογίες, ίσως να πρέπει να σας πω κάπως έτσι Μην ε, κάνετε και τόσες πολλές τροπολογίες. Αλλά βεβαίως να υποβάλλετε τις σημαντικές τροπολογίες. Και λοιπόν, περιμένοντας τις τροπολογίες σας, υπάρχουν ακόμα κάποια πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν. Και ναι, περιμένω. Τις περιμένω, μετά θα τις συζητήσουμε και θα φτιάξουμε μια καλή έκθεση που ελπίζω ότι θα θεωρηθεί ότι στηρίζει την πορεία. Αν και επικρίνει τα όσα δεν λειτουργούν, γιατί σε μια φιλία πρέπει κανείς να ισχύει κριτική γιατί διαφορετικά δεν λειτουργεί η φιλική αυτή σχέση. Ευχαριστώ πολύ. Να θυμίσω ότι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών θα είναι το ίδιο όπως για την Τουρκία 18 Ιανουαρίου το στις 12 το μεσημέρι. Και περνάμε στο τελευταίο σημείο για σήμερα που είναι η, συζήτηση των νομοθετήσεων της ΑΦΕΤ για την έγκριση της διαχείρισης από πλευρά της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για το 2015. Δύο νομοθετήσεις έχουμε και ε, αρχικά να πω ότι όσον αφορά την έγκριση της ε, δημοσιονομικής διαχείρισης στην ΑΦΕΤ έχουμε να αντιμετωπίσουμε το, να εξετάσουμε μάλλον πώς ε, διαπανώνται τα χρήματα και να αποφύγουμε τις ε, σπατάλες ε, φυσικά λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα των εξωτερικών δράσεων. Γι' αυτό χαίρομαι που φαίνεται να υπήρχε σημαντική ισορροπία. Στην περίπτωση της διαχείρισης ε, του κτηρίου, για παράδειγμα, της, εξωτερικής εξωτερική της υπηρεσίας εξωτερικής είναι ένα θέμα που αντιμετωπίσαμε και πέρσι και έχουμε πραγματικά προβλήματα που εντοπίσαμε και πρέπει να τα προσεγγίσουμε. Όμως δεν θα πρέπει να, χάσουμε, να ξεχάσουμε ούτε να γνωρίσουμε τα το γεγονός ότι 139 είναι οι χώρες που υπάρχει αποστολή μας ε, και όπου ε, λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε και την υπεραντιπροσώπευση των εθνικών μας εκπρόσωπων ε, σε συγκεκριμένους τομείς των διαφόρων μάλλον εθνικοτήτων στις διάφορες υπηρεσίες της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και τώρα θα πρέπει να δώσω το λόγο στον κύριο Λίτζη που θα μιλήσει εξ ονόματος του εισηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως είπατε, εγώ θα σας διαβάσω δύο την εισήγηση του κυρίου Μπαλσίτη. Θέλω να παρουσιάσω τις βασικές γραμμές της γνωμοδότησης όσον αφορά την απαλλαγή της Κομισιόν και της, των εκτελεστικών υπηρεσιών της για το, την οικονομική χρήση 2015. Τονίζεται ότι δυστυχώς το επίπεδο σφάλματος στο τίτλο 4 για το 2015 όπως έχει εκτιμηθεί από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια του έκθεση δεν έχει μειωθεί το περιθώριο αυτό σφάλματο σε σχέση με το 2014 και ανέρχεται σε 2,8%. Δεύτερον, ωστόσο, αυτό είναι κάτω από το επίπεδο αποδεκτού και εντοπισμένου σφάλματος σε άλλου τίτλους, ε, παρά το γεγονός ότι ε, οι δραστηριότητες της Ένωσης Εξωτερικής ε, Δράσης συνήθως γίνεται σε ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον. Τέταρτον, στηρίζοντας τις συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου, ε, καλωσορίζουμε το γεγονό ότι η Κομισιόν έχει πλήρω εφαρμόσει πέντε από τι εφτά συστάσει που είχε υποβάλει το Ελεγκτικό Συνέδριο το 2012 και το 2013 μέσω των εκθέσεών του. Επίση, παροτρύνουμε την Επιτροπή να λάβει μέτρα ώστε να ολοκληρώσει την εφαρμογή των δύο υπολοιπωμένων συστάσεων. Ο κ. Μπαλσίτη κατέθεσε δύο επιπλέον τροπολογίε για να συμπληρώσει τη γνωμοδότηση που σχετίζεται με τις αποστολές του CSPD. Ε, Επίση, ε, για τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν για το τμήμα 3 και για τις νέες παραγράφους 6α ε, και 6β, ο κύριος Βαλθίτης τι καλωσορίζει γιατί συμπληρώνω θετικά αυτή την έκθεση. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μακάλιστερ, εξ ονόματος του κύριου Πρέντα. Yes, Chair. Thank you very much. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ και εξ ονόματο του κυρίου Πρέντα, ο οποίο δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί σήμερα, θα ήθελα να σα διαβάσω την εξή δήλωση. Θα ήθελα καταρχά να ζητήσω συγγνώμη που δεν μπορώ να παρευρεθώ σήμερα εδώ για το θέμα τη απαλλαγή του 2015. Να ευχαριστήσω ύστερα τον εισηγητή για το σχέδιο τη έκθεση. Κατέθεσα μόνο λίγες τροπολογίες σε ό,τι αφορά το σχέδιο του προπολογισμού, θα ήθελα να αναφέρουμε το δικαστήριο, το ελεκτικό συνεδρίο και την έκθεση του για την ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων στα Δυτικά Βαλκάνια. Γι' αυτό λοιπόν και καλώς ορίζουμε για τις στάσεις του ΙΣΥΕ προς την κατεύθυνση αυτή. Σε ό,τι αφορά επίσης την ενίσχυση ε, τις ε, που παρέχεται προ τι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων και στην τροπολογία 20 αναφέρεται η παροχή βοήθεια προ τη Μολδαβία και την Ουκρανία και γίνεται πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει χρήση τη μόχλευση προ τι χώρε αυτέ για να υπάρχει και σωστή παρακολούθηση τη των ε, μεταρρυθμίσεων που γίνονται. Και επίσης ε, θεωρώ ότι αυτές οι δύο τροπολογίες έχουν να κάνουν πολύ σημαντικά θέματα. Ελπίζω λοιπόν να τις υποστηρίξει η Επιτροπή μας σε ό,τι αφορά το σχέδιο έκθεσης για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Να σας πω ότι κατέθεσα μόνο δύο μικρές τροπολογίες σε ό,τι αφορά την σωστή εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροπολογία 4 για τη σωστή εκπαίδευση του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 14 υποστήριξη για την σωστή διαχείριση των κτίριων. Προσβλέπω στη συζήτηση των σκιωδών εισηγητών και στα σχόλια όλων και στην γενικότερη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταρχάς ο κύριος Ρωμαν Μακαγκούσταρ από την Υπηρεσία Εξωτερικής Πολιτικής Δράσης. Ευχαριστώ, πολύ. πολύ. Για το σημείο 5 του σχεδίου γνώμοδότησης θέλουμε να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι οι αποστολές της ΚΕΠΑ και ο λογιστικός έλεγχος των αποστολών αυτών για να συνάδουν με το άρθρο 60 του Δημοσιονομικού Κανονισμού είναι χρονοβόρες διαδικασίες λόγω της πολυπλοκότητος και του πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργούν αυτές οι αποστολές. Μέχρι στιγμής έχουμε τέσσερις τέτοιες αποστολές βάσει του άρθρου 60 και είναι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της ΚΕΠΑ, η ΟΥΛΕΞ Κόσοβο, η ΟΥΠΟΛ Αφγανιστάν, η ΟΕΜ Γεωργία και η στην Παλαιστίνη. Συνεχίζεται το έργο για την συμμόρφωση σε σχέση με την ΕΟΚΑΠ στο Νίγηρα και η και σε σχέση με τις ε, υπολοιπόμενες αποστολές η UMRAFA, η Ukraine και Μάλι ε, έχουν, είναι στο στάδιο της εκκίνησης, είναι έτοιμες να κινήσουν και για την αποστολή με τη Λιβύη δεν είναι δυνατόν λόγω των επιτοπίων συνθηκών να, να έχουμε μια πραγματική αξιολόγηση για αυτή την έκθεση, για την αποστολή. Σας λέω και πάλι ότι είναι έργο εν εξελίξη όλα αυτά και ο στόχος μας είναι να τηρήσουμε την σύσταση του ελεκτικού συνεδρίου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ενρίκε Γαρσία από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Εκτιμούμε την εξισορροπημένη παρουσίαση του εισηγητή για το θέμα της ε, απαλλαγής. Συμφωνούμε με την παρουσίαση αυτή. Εξακολουθεί να υπάρχει ένα επίπεδο σφαλμάτων, αλλά αναγνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο το περιβάλλον στο οποίο πρέπει να λειτουργήσουμε και αυτό οδηγεί σε ένα επίπεδο σφαλμάτων το οποίο παρόλα αυτά είναι χαμηλότερο από ό,τι σε άλλους τομείς πολιτικής. Ακόμα και αν είμαστε πάνω από το 2% νομίζουμε ότι πηγαίνουμε προς σωστή κατεύθυνση Έχουμε καλές λοιπόν ενδείξεις προς την κατεύθυνση αυτή. Έχει μειωθεί το ε, σφάλμα το οποίο είναι το ε, σφάλμα από τα 4 στα 2% και ελπίζουμε ότι καλά τα πάμε. Μας ικανοποιεί επίση και η θετική αξιολόγηση του ελεκτικού συνεδρίου σε σχέση με την εφαρμογή των συστάσεών τους από τα προηγούμενα έτη Όπω ξέρετε είναι πολύ σημαντικέ αυτέ οι συστάσει για την ενίσχυση του ελεκτικού μα συστήματο, και γι' αυτό έχουμε συμφωνήσει με όλε αυτέ τι συστάσει εφέτο και είμαστε ευτυχισμένοι γιατί το δικαστήριο έχει αξιολογήσει θετικά το έργο μας για την εφαρμογή αυτών των συστάσεων. Οι περισσότερες από αυτές μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν εφαρμοστεί πλήρως και μία έχει εφαρμοστεί στα μεγαλύτερα σε, σε γενικές γραμμές για τις ε, επαληθεύσεις σε σχέση με τους τελικούς ε, δικαιούχους. Συνεργαζόμαστε με το ελεκτικό συνέδριο και έχουμε κάνει τα απαραίτητα μέτρα και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι θεωρούνται ότι έχουν εφαρμοστεί οι συστάσεις στο μεγαλύτερο βαθμό τους και αυτή τη στιγμή αλλά εξετάζουμε την ε, αναθεώρηση των όρων αναφοράς για το λογιστικό έλεγχο επί τη βάση κριτηρίων που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τα ασφάλματα τα οποία υπάρχουν σε αυτές τις ε, συναλλαγές. Κατά τα άλλα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον συναδελφό μου την Digenia. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο μήνους από την Digenia. Ε, Ευχαριστώ, αξιότιμοι βουλευτέ, και θα πρέπει να σα πω ότι χαιρόμαστε ιδιαίτερα για το γεγονό ότι μα δίνει την ευκαιρία να διευκρινίσουμε την κατάσταση σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο περιθώριο σφάλματο για το 2015. Θα ήθελα να τονίσω καταρχά ότι το θέμα αυτό έχει να κάνει με, ένα συγκεκριμένο τρόπο διαχείριση ή έμεση διαχείριση με την χώρα δικαιούχου που έχει να κάνει με το ΙΠΑ, ε, δηλαδή την, ε, το μέσο το προενταξιακό. Το 2015 λοιπόν εντοπίζονται ε, αδυναμίες σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό και θα πρέπει να σας πούμε ότι τα συμπεράσματα γίνονται βάσει της ε, αντιπροσωπευτικότητας του συντελεστή αυτού σφάλματος και θα πρέπει να σας πούμε ότι στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής ε, περιλαμβάνονται διάφορα τέτοια στοιχεία για την ε, έκθεση ετήσιας δράση το 2015. Έχουν λήφθει υπόψη πλήρω οι συστάσει του Ελληνικού Συνεδρίου για τον υπολογισμό του υπολοιπόμενου συντελεστή ε, σφάλματος για το τμήμα των ε, δικαιούχων, των ε, χωρών που λαμβάνουν επιδότηση. Άρα κάναμε δύο πράγματα. Ενισχύσαμε τις δραστηριότητές μας και αναπτύξαμε ένα σχέδιο δράση. Και αυτά τα μέτρα λοιπόν λάβαμε στα πλαίσια του σχεδίου δράση. Καταρχά, τα υφιστάμενε συμβάσει άρια που καλύπτουν το ΙΕΝΑΙ e προ το παρόν, δηλαδή το μέσο γειτονία σε όλα τα τμήματα διαχείριση και την ΑΙΠΑ, έμεση και άμεση διαχείριση, καλύπτει πλέον και την ΑΙΠΑ και το INBC2. Κατά δεύτερον, Τρεις έλεγχοι έχουν γίνει από την DJ στην Κροατία, στην Τουρκία και στην πρώην Δημοκρατία της Μακεδονίας που συνδυάζουν την εκ νέου χρήση των ελέγχων και ελέγχους ε, αποδόσεις. Και κατά τρίτον θα πρέπει να σας πούμε ότι δόθηκε εντολή σε εξωτερικούς ε, ελεγκτές για να γίνουν επιπλέον έλεγχοι στην Τουρκία και στην Πουγουμουδού σε μεγαλύτερο τμήμα των συναλλαγών για να υπολογιστεί καλύτερα ο συντελεστή σφάλματο. Να σα υπενθυμίσω ότι για την ακρόαση του Επιτρόπου Χαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στι 8 Νοεμβρίου πέρσι, η κυρία Λαμάρκα από το ελεκτικό συνέδριο ανέφερε ότι το ελεκτικό συνέδριο είναι ικανοποιημένο με τις δράσεις που προτείνονται από την DGNIR και ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα φροντίσουν να υπάρχει καλύτερη αξιοπιστία και αντιπροσωπευτικότητα του υπολοιπόμενου συντελεστή εισφάλματος του 2015 και ότι έτσι θα δώσουμε απάντηση σε όλα τα σημεία κριτικής τα οποία απεύθυνε το ελεκτικό συνέδριο. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Πατρίσια Ρεμπούσκα από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ τους αξιότιμους κύριους βουλευτές ε, για τη σημερινή συνεδρίαση και επειδή μας δώσατε την ευκαιρία να έρθαμε και να συζητήσουμε μαζί σας σήμερα. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην απαλλαγή και στις γνωμοδοτήσεις που συντάσσουν οι διάφορες επιτροπές, ιδιαίτερα καθώς η ΑΦΕΤ παρακολουθεί στενά τη συμβολή του κοινοβου, της Ένωσης στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Είναι πολύ καλή ευκαιρία για μας να αξιολογήσουμε και να κατανοήσουμε που χρειάζεται να υπάρξουν βελτιώσεις, να δείξουμε και να συσκετήσουμε την προσήλωσή μας στις χρηστές οικονομικές προεπτικές αλλά και να δούμε τι επέτυχε ε, το θεσμικό μας ή ε, το θεσμός μας και πάλι είμαι ευτυχής που μπορώ να πω ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, μπορεί να δείξει χαμηλό ποσοστό σπάρματος κάτω από το 2%. Αυτό για ένα νέο θεσμό όπως ο δικός μας είναι σημαντικό επίτευγμα που θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε και να στοχεύουμε και στα επόμενα χρόνια. Το ελεγκτικό συνέδριο έχει αναφέρει βασικά δύο ανησυχίες και έχει κάνει δύο συστάσεις σε σχέση με την πρόσληψη των αντιπροσωπιών για τις τοπικές υπηρεσίες. Είναι πολύ δύσκολο γιατί κάποιες φορές έχουμε 300 ανθρώπους για, που, ζητούν, που, που, που, που αίτηση για τη θέση του οδηγού και θα πρέπει να αποκολουθούμε αυτές τις διαδικασίες με ισορροπημένο τρόπο σε αυτό το τομέα. Χωρίς... Τώρα, όσον αφορά τις προμήθειες, ε, ε, η υπηρεσία εξωτερική δράση ε, πέρσι το 2014 ήταν πολύ σημαντικό στασμός. Μελετήθηκαν 500 διαφορετικές, 50 συγγνώμη, διαφορετικές συναλλαγές για προμήθειες και το συνέδριο είπε ότι αυτές οι διαδικασίες είναι πολύ ψηλής ποιότητας, πάνω από το 135 ή 137%. Δεν έγιναν παρατηρήσεις καν και οι παρατηρήσεις του ελληνικού συνεδρίου εστιαστήκαν στις διαδικασίες μέσης και χαμηλής αξίας και τα λαμβάνουμε πολύ σοβαρά αυτά υπόψη και θα τα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια. Έχουμε προκλήσεις, έχουμε 139 αντιπροσωπείες αποκεντρωμένες σε 139 ε, διοικήσεις και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε στο μέλλον. Οι παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη και όπως είπατε στο πλαίσιο του, της διαδικασίας για τον προπολογισμό του 17 έχουμε ε, συμφωνήσει με το Κοινοβούλιο για την πετώπιση θέματων ε, προσωπικού, ιδιαίτερα την ισορροπία ανάμεσα στις, ε, στην, εκπροσώπηση των διαφόρων κρατών μελών όπου υπάρχουν ανισορροπίες. Να θυμίσουμε ότι το ποσοστό παρουσίας διπλωματών από τα κράτη-μέλη στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης αντιστοιχεί σε αυτό που θεσπίζεται από τον νομικό πράξη που θεσπίζει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Όμως, όπως αναγνωρίζετε, υπάρχει κάποια ανισορροπία όσον αφορά την εκπροσώπηση στους επικεφαλείς των αντιπροσωπιών με καλύτερη παρουσία διπλωματών των κρατών μελών, ενώ όταν βλέπουμε την μέση, το, την μέση, τα μεσαία στελέχη ε, αντιστρέφεται η κατάσταση. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα, ενώ έχουμε και την ε, διαδικασία κινητικότητας και βεβαίως εφόσον επικρατεί ε, ε, αξιοκρατία. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλε προκλήσει στην υπηρεσία εξωτερική δράση, γιατί όπω είπα στην αρχή, ήμασταν ένα μικρό θεσμό, αλλά τελευταία έχουμε μετατραπεί σε πολύ μεγάλη, ε, με σημαντικό θεσμό και έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλα και περισσότερες προκλήσεις με όλα και λιγότερους πόρους και σε πολύ δύσκολο περιβάλλον όσον αφορά την ασφάλεια και αυτό είναι μεγάλη μας ανησυχία να έχουμε την απαραίτητη ασφάλεια για τις αντιπροσωπείες μας και θέλω με αυτή την ευκαιρία να σας ζητήσω μάλλον να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για τη στήριξή του για το προϋπολογισμό του 2017 όσον αφορά την ενίσχυση του προσωπικού ασφαλείας στις αντιπροσωπείες μας. Ίσως να χρειαστούμε να επανέλθουμε για αυτό το θέμα. Και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και εκ των υστέρων για όλη την στήριξη που μας έχετε προσφέρει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να θυμίσω ότι η ψηφοφορία για αυτές τις νομοδοτήσεις θα γίνουν στις 31 Ιανουαρίου 2017 και έτσι ολοκληρώνεται η απόψηνή μας συνεδρίαση. Η επόμενη θα γίνει στις 24 Ιανουαρίου εδώ στις Βρυξέλλες. Αντίο σας.